Good afternoon, colleagues. We begin with the adoption. Καλησπέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινούμε με την έγκριση τη ημερησία διατάξεω. Επίση, έχω να σα πω για κάποιε αλλαγέ στο σχέδιο τη διατάξεω για το σημείο 6, το οποίο είναι η, το σχέδιο έκθεση για λειτουργία του χώρου Σέγγεν. Ο εισηγητή Καλός Κοέλιο ανέβαλε την παρουσίαση για την 8η Μαρτίου στη συνεδρίασή μα. Όταν λοιπόν, έχετε κάποια ένσταση, εγκρίνουμε την. Ε, σε διάταξη έχουμε, ε, δυστυχώς δεν έχουμε κροατικά και ιρλανδικά και ελτικά τέλο πάντων και επίσης συγκρίναμε την καινούργια κατησόδοξη πράξη 26 Δευτέρου 18 όσον αφορά κάποιες πρόδρομες φαρμακευτικές ουσίες όσον αφορά κάποια λίστα ε, προγραμματισμένων όπως μας ουσιών και υπάρχει μία προθεσμία 2 τρίτου ε, μόνο δύο τρίτου λάβατε τα, τα σχετικά και σε δύο μήνες μπορεί σχετικά με αυτά να υποβαλήσετε στο Κοινοβούλιο. Επίσης, για την συλλογή δεδομένων των κρατών μελών για στατιστικέ δεδομένα όσον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος εισόδου-εξόδου για την εφαρμογή του νόμου. αυτή είναι μια εφαρμοστική απόφαση. Επίσης, αν υπάρχει κάποια ένσταση σχετική η προθεσμία, θα πρέπει να υποβληθεί στη γραμματεία μας πριν τις 16 Τρίτου του 18. Έγινε στο πρωτικό για 15 Έκτου. If there no objections to the minutes. Αν δεν έχετε στάση για τα πρακτικά, τότε αυτά εγκρίνονται. Και τώρα θα φτάνουμε στο σημείο υπαριθμών 4. Είναι από τα βασικά σημεία σύντησης για σήμερα και Καλώς ήρθαμε την κυρία Γιάλα Σέντερ, η οποία θα συμμετάσχει σε αυτή την συζήτηση για αυτή την κοινή συνεδρίαση με την Τροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Είναι επίσης πρόεδρος της Συνεπροσωπής για σχέση με τις χώρες του Μαγρέμπ και ε, ε, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών ε, Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, ο κύριος Περμούη. Και οι δύο καλώ όρισαν στην Επιτροπή μα, στην Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, συνάδελφε, και αφορά την τρέχουσα κατάσταση στην Λιβύη. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμο το ότι αυτά τα κάνουμε σε μια κοινή συζήτηση. Πρόσφατα προτείναμε να κάνουμε μια αποστολή στην ε, περιοχή του Μαγρέμπ και πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η ενημέρωση. Επίσης έχουμε συνοηθεί και με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης που εκπροσωπείται σήμερα στην συζήτησή μας. δώσουμε το λόγο στην κυρία Σέντερ, αλλά κατόπιν και στον κύριο Πέρμουι για κάποιες ε, προεισαγωγικές σύντομες παρατηρήσεις για να δώσουν το ανακτήριο λάθισμα ή στην συζήτηση. Όχι, όμως μου είπανε ότι πρώτος θα μιλήσει ο κύριος ε, Περμουή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Έχετε το λόγο. Να σας τα πω στα ισπανικά λέω κύριε Περμουή. Σα ευχαριστώ πρώτα σε αυτή την ε, ευκαιρία εδώ να μιλήσουμε με την φορέα αυτό των ε, Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά για το τι γίνεται στη Λιβύη αλλά και, σε, και αλλού στον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το, επίσης το ότι πρόκειται σε όλα αυτά να συνεργαστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τον Νοέμβριο πέρσι ήταν πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία μας για να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει με την δραματική κατάσταση των ε, προσφύγων μεταναστών στην ε, Λιβύη. Είχαμε πάνω από 9.000 που επέστρεψαν στη χώρα ε, Προέλευση και 200 οι οποίοι ζήτησαν άσυλο, αλλά οι τους με μετακίνηση από την ε, Λιβύη. Άρα είναι βελτίωση. Όμως έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους πρόσφυγες μεταναστές που ζουν στη Λιβύη πάρα πολύ, σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και πάρα πολλοί αυτούς είναι κλεισμένοι σε κάποια κέντρα κράτησης και διαμονής τέλο πάντων. Οπότε θα πρέπει οι προσπάθειες να ενταθούν ούτως ώστε να βοηθήσουμε όσους χρειάζονται την διεθνή ε, βοήθεια. Επίσης θα πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα τι θα γίνει, πώς θα μπορέσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες για να μπορέσουμε να πετύχουμε μια πολιτική και βιώσιμη λύση στην ε, λιβική κρίση. Επίσης ε, είναι σημαντικές προσπάθειες του ΟΗΕ για μια διαδικασία πολιτική στο πλάι της ε, Λιβύης και Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις. Είμαστε με τον ειδικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματείου το ΙΕ του τον ε, Διαστάρ Σαλαμέ σε ζητενή επαφή για να μπορέσουμε να δούμε πότε θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια συνάντηση, κάποια συζήτηση. Τέλος, ο, ο συνάδελφος Παντζέρη ε, των σοσιαλδημοκρατών δεν μπόρεσε σήμερα να έρθει στην συνάντηση. Πάντως έχει ένα κείμενο ε, σχέδιο σύστασης προς ε, το Συμβούλιο και την Κομισιόν για την Λιβύη. Και στις 23 Τετάρτου πρέπει να το συζητήσουμε και στις 24 ε, Απριλίου πρέπει να γίνει η έγκριση του σχετικού κειμένου της ε, σύστασης αυτής. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Αγιάλα Σέντερ. Σας ευχαριστώ κύριε Περμού, ευχαριστώ και εσάς κύριε Πρόεδρε και εγώ να ε, καλωσορίσω τον εκπρόσωπο της είπα της του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε αυτή την ε, κοινή συνάντηση και όπως και ο κύριος Κόουσο θέλω να πω ότι βοηθούμε όσο μπορούμε περισσότερο τη δραστηριότητα του ΟΗΕ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η υπόθεση γιατί η Λιβύη είναι μια χώρα που μας προβληματίζει πάρα πολύ και επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι πρέπει από το χέρι μας και όλα αυτά τα κάνουμε από κοινού με τον ε, ΟΗΕ για την χώρα εκείνη. Και όλα αυτά να γίνονται με έναν τρόπο ολοκληρωμένο, σφαιρικό για όλη τη χώρα, λαμβάνοντα υπόψη το παρελθόν, αλλά και το μέλλον αυτής της χώρας. Και βεβαίως θα πρέπει να ε, εξετάζουμε καμιά φορά όμως τη χώρα σε κάποιο είδους κατάτμιση κομμάτι-κομμάτι αλλά θα πρέπει φυσικά το σύνολο του οράματός μας, της άποψή μας, της έποψής μας στον κόσμο να είναι συνολικό και στις 25 Ιανουαρίου τα είπαμε και ως ε, διακοινωτική επιτροπή με το Μαγρέμπ ανταλλάξαμε απόψεις αλλά και με τον κύριο Πικέ ε, της εξωτερικής ε, υπηρεσίας και με τον κύριο Λαουίν από την Λιβύη και στην συνάντηση εκείνη ε, υπήρξαν κάποια νέα που είναι θετικά και έτσι βαθμία έχουμε αυτούς τους εκτοπισμένους στο ιστορικό της χώρας και αυτοί έχουν πρόβλημα αλλά είπαμε ότι κατά όλους μεγάλες προσπάθειες από την ΑΚΝΟΡ και επίσης από διάφορες ΜΚΟ και από τον ΟΗΕ να επιστρέφουν κάποιοι από αυτούς στις πόλεις ε, καταγωγής τους. Επίσης βοηθούμε με ενέργειες πρόληψης, ε, προσπαθούμε να κάνουμε κάποιο είδους ναρκαλίευση, ε, εντοπισμό κλπ. Οπότε υπάρχει αυτή η αποστολή υψηλού επίπεδου της Αφρικανικής Ένωσης εκεί του ΟΗΕ και, του, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τρίπολη στις 22 Φεβρουαρίου. Εκεί πρόκεισαν κάποια σημαντικά στοιχεία για το πώς είναι δυνατόν να μπορέσουμε να βαθμίσουμε τη συνεργασία μας με τις Λιβυγές Αρχές και έτσι να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε μια καλύτερη ε, ε, αντίδραση σε όλα αυτά τα προβλήματα. Α, γι' αυτό λοιπόν και περιμένουμε πώς και πώς να ακούσουμε τι έχει να πει ο κύριος Πικέ και ο κύριος Μορντή για αυτά τα αποτελέσματα. Ε, των ενεργειών και επίσης να σας ενημερώσω ότι η διάσκεψη των Προέδρων επεκύρωσε το ότι θα πρέπει να γίνει μια αποστολή ad hoc στην ε, Λιβύη το συντομότερο δυνατόν μια από τις τελευταίες εβδομάδες υπήρχαν προβλήματα σε επίπεδο ασφάλειας οπότε θα πρέπει να έχουμε πρόεδρο της αποστολής την ε, πρόεδρο τη ε, Διακοινωνικής Επιτροπή, αλλά και του πρόεδρους των Σερμοδίων Επιτροπών τη ΑΦΕ, δηλαδή τη ΛΥΜΠΕ και της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οπότε προπαρασκευόμαστε για αυτή την τόσο σημαντική αποστολή και μόλι έχουμε κάτι συγκεκριμένο πρόκειται να σα ενημερώσουμε. Και σα ευχαριστώ. Ο Πρόεδρο, σα ευχαριστώ και του δύο. Και τώρα, το λέγει και Καρμέν Σάκερ, φαλής της ε, μονάδας για την Βόρεια Αφρική. Η κυρία Σάκαρ, να μας ενημερώσει για το έργο της στην Λιβύη. Thank you very much for inviting Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Θα έχουμε την ευκαιρία να εξηγήσουμε λίγο περισσότερο τι κάνει η Αρμοστία στη Λιβύη και ποιες είναι οι προτεραιότητές μας και πώς έχουμε οργανώσει τις παρεμβάσεις μας. Να εξηγήσω πρώτα απ' όλα ποιε είναι οι προτεραιότητέ μα ε, στη Λιβύη. Είναι τέσσερι οι τομεί που μα απασχολούν. Ε, ενίσχυση των σχέσεων με τι αρχέ τη Λιβύη για να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κατάσταση της χώρας. Προσπαθούμε να επεκτείνουμε τα προγράμματά μας. Είναι μια χώρα που διαρκώς μεταβάλλεται η κατάσταση ακόμη και εκεί που έχουμε περιορισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση. Ασχολούμαστε με τους ιστορικούς εκτοπισμένους πληθυσμούς, τις κοινότητες υποδοχής και αυτούς που επιστρέφουν από από εκτοπισμένους πληθυσμούς. Κοιτάζουμε να προσφέρουμε βοήθεια σε πρόσφυγες και τον τεσσάσυλο. Θα περάσω σε λεπτομέρειες για κάθε μια από αυτές τις ομάδες, αλλά είναι σημαντικό να πω ότι η Λιβύη δεν είναι η πιο εύκολη χώρα όπου μπορούμε να εκτυπλώσουμε τις δραστηριότητές μας. Η κατάσταση της ασφάλειας είναι αμφιρόπη και με τη, χώρα, με ασχολούμαστε τα τελευταία 27 χρόνια, από το 1991, από το 2014, τον Ιούλιο του 2014, όλο το σύστημα του ΟΗΕ λειτουργεί με βάση την, ε, την Ισία, αυτή είναι η έδρα μας προς τη Λιβύη. Δεν εγκαταλείψαμε ποτέ τη Λιβύη, συνεχίζουμε να έχουμε παρουσία μέσω του προσωπικού μας επιτόπου στην Τρίπολη και τη Βεγγάζη, αλλά από το 2016 συστηματικά Στέλνουμε και ξένους συνεργάτες σε αποστολές και συνεχίζουμε τις δραστηριότητές μας για την καταγραφή, την εκμερίωση και την ταυτοποίηση των ευάλωτων ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασία. Ο πληθυσμός που μας απασχολεί κυρίως είναι 500 και περίπου 15.000 άτομα που χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Τους εσωτερικώς εκτοπισμένους, 180.000 τους ε, επιστρέφοντες, περίπου 314.000 και μετά έχουμε 40.000 ε, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. 50.000 το σύνολο. Από το 2016 η Αρμοστία έχει καταγράψει 10.000 αιτήσει ασύλου παρά τις δυσκολίες ε, με την ασφάλεια και τις ε, εντολές εκένωσης που είχαν δοθεί ακόμη και στους συνεργάτες του ΟΗΕ. Μια από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε στη χώρα ήταν οι περιορισμοί σε ό,τι αφορά τις ε, υπηκότητες, τις ηθαγένειες. Η ύπατη αρμοστία ζητήθηκε να ασχοληθεί με 7 και αν δεν τις γνωρίζετε, μιλάμε για Σομαλία, Σουδάν, Ερυθρέα, Αιθιοπία, Συρία, Ιράκ, Ιράκ και Παλαιστίνη παρά τον περιορισμό συστηματικά ε, είχαμε συζητήσεις με τις αρχές της Λιβύης και πρόσφατα είχαμε και τη δυνατότητα να λάβουμε μερίμνα για την Ιεμένη και τους Σαουδάραβες που, και τη Σαουδική Αραβία και τους πολίτες τους. Έχουμε αυξήσει τα κονδύλια μας και τις περιοχές παρέμβασης ιδίως με τη Σαμπράτα και την Ταουέργα πιο πρόσφατα. Κοιτάξαμε και προσφέραμε βοήθεια τουλάχιστον σε 1.200 ε, άτομα, 300-400 οικογένειες που ήθελαν να επιστρέψουν στην πόλη τους με την Ταουάργα, αλλά δεν μπορούσαν λόγω των εχθροπραξιών. 50 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά της ε, Ταουάργα και κοντά στη Σύρτη. Κοιτάξαμε να τους προσφέρουμε τρόφιμα, σκηνές, νερό και ένδυση για το χειμώνα και σχεδιάζουμε το 2018 να εφαρμόσουμε 200 quip, όπως λέγονται, ε, σχέδια γρήγορης αντίδρασης που θα ωφελήσουν και τις κοινότητες ε, υποδοχής των εσωτερικών εκτοπισμένων και τις ε, κοινότητες των προσφύγων για να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων για τους πρόσφυγες και τους ετούντες άσυλο συνεργαζόμαστε με το Διεθνή Οργανισμό για τη Μετανάστευση στη μεικτή ομάδα για τους πρόσφυγες. Έχουμε 12 σημεία ε, καταγραφής μαζί με τους ε, συνεργάτες μας για να προσφέρουμε συνδρομή. Υπάρχουν 6 ε, σημεία αποβίβασης όπου συνεργαζόμαστε με τον Οργανισμό Μετανάστευση και συνεργαζόμαστε και με την ακτοφυλακή τη Λιβύη για όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικοδόμηση δυνατοτήτων, ταυτοποίηση και την ε, αναπομπή των αιτήσεων ανθρώπων που χρειάζονται διεθνή προστασία. Για τον ε, πήγοντα μηχανισμό μετάβασης που έχει αρχίσει να λειτουργεί από τον Νοέμβριο, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι από τον περσινό Νοέμβριο οι περισσότερες από τις αποφάσεις των λιβικών αρχών να απελευθερώσουν ανθρώπους από τις φυλακές είχαν να κάνουν ε, με την ανάγκη να εκενωθούν κάποιες περιοχές. Η υπατηρεμοστία λοιπόν έχει προβλέψει ένα μηχανισμό της ε, κατεπίγουσας διέλευσης, διαμετακόμισης των ανθρώπων που είναι πλέον βάλλοντα ε, και πρέπει να φύγουν από τα κέντρα κράτησης στον Ήγηρα. Μέχρι τώρα έχουν φύγει 1.334 προσφύγες και τον από αυτά τα κέντρα οι 1020 έχουν ε, ανατεθεί στην κυβέρνηση του Νιγήρα που ήταν ε, πολύ ανοιχτή, συνεργάσιμη και φιλόξενη και 312 μεταφέρθηκαν απευθείας στην Ιταλία όπου η κυβέρνηση έχει αναλάβει την ευθύνη για την προστασία τους ως προς το καθεστώς του πρόσφυγα. Ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να τονίσουμε είναι οι δυσχερείς συνθήκες, οι συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν στα κέντρα <coughs> κράτησης και στις εγκαταστάσεις. Δεν υπάρχουν επαρκείς συνθήκες υγιεινής, ε, δεν υπάρχει δυνατότητα συμβουλευτικής, δεν υπάρχει ιδιωτικότητα στις συνεντεύξεις, και πέραν όλων αυτών η Πατιαρμοστία κάνει ό,τι μπορεί για να τους καταγράψει και να εντοπίσει τους πλέον ευάλωτους για να τους ε, μεταφέρει αλλού. Για την ε, επαναγκατάσταση είναι σημαντικό να τονίσουμε την ανάγκη περισσότερης διεθνούς αλληλεγγύης σε ό,τι αφορά τις ποσοστώσεις. Προσπαθούμε να συνεννοηθούμε με την κυβέρνηση τη Λιβύης για του πλέον ευάλωτου, αλλά μόλι απελευθερωθούν από τα κέντρα κράτηση πρέπει να του βρούμε κάποια λύση. Αυτό επιδιώκουμε και αναζητούμε νομικές οδούς, νομικούς διάβλους και τις ποσοστώσεις μετεγκατάστασης. Τον Δεκέμβριο του 2017 είπα η αυτή απίφθηνε έκκληση για 1.300 θέσεις μετεγκατάστασης για την ομάδα αυτή των 1300 που είχαμε κενώσει με τον μηχανισμό κατεπίγουσας ε, διαμετακόμισης προς τον Ήγηρα. Ως τώρα έχουμε λάβει 1100 ε, θέσεις, υπάρχει δέσμευση για τόσες θέσεις, εκ των οποίων κάποιες είναι από ευρωπαϊκέ χώρε και αυτό το εκτιμούμε πολύ. Χρειάζεται όμω να προβλεφθούν περισσότερε θέσει και να επιδειχθεί περισσότερη αλληλεγγύη. Εάν θέλουμε να μετεγκαταστήσουμε 5.000 έως 10.000 πρόσφυγες, εμείς μπορούμε να ασχοληθούμε με την ταυτοποίηση και τις συγκεκριμένε υποθέσεις. Όμως πρέπει και οι χώρες λιγάκι να προταθούν και να ασχοληθούν με τις υποθέσεις. Ο Νίγηρας ως τώρα έχει παραλάβει 1.020. Μόνο όμως 25 άτομα έφυγαν ε, προς τη Γαλλία μετά τις συνεντεύξεις τους. Πρέπει να φύγουν περισσότεροι από τον Ήγηρα, διότι ιδάλλως δεν θα μπορέσουμε να στείλουμε περισσότερους ανθρώπους από τη Λιβύη. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να δείξουν οι κυβερνήσεις ότι είναι συνεργάσιμες, ότι μπορούν να εκφράσουν αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες. Και η διεθνής κοινότητα ότι μπορεί να αναλάβει την ευθύνη. Τέλος, πολύ σημαντικό επίσης, να πούμε πόσο σημαντικό είναι η υπατιαρμοστία να συνεχίσει να έχει πρόσβαση όχι μόνο στις 7 ηθαγένειες και τις πλέον δύο που σας ανέφερα, ε, με τις οποίες εργαζόμαστε στη Λιβύη, αλλά σε όλους που έχουν ανάγκη από διεθνή προστασία. Ο Διεθνής Οργανισμός ε, ασχολείται με την ε, εκένωση, με την διαμετακόμιση ανθρώπων από τα κέντρα κράτησης, αλλά έχουμε περιοριστεί σε κάποιες ηθαγένειες υποτίθεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι που βρίσκονται σε κράτηση δεν θα τους ε, κοιτάξουμε, αλλά για αυτούς προέρχονται τη λαϊκή δημοκρατία του Κογκό, από την κεντροαφρικανική δημοκρατία ή άλλες εφαγένειες. Μπορεί να μην χρειάζονται διεθνή προστασία, ε, έχουν όμως άλλες ανάγκες. Δεν σημαίνει ότι όλοι χρειάζονται την ίδια ακριβώ βοήθεια συνδρομή. Παρ' όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν ε, οι κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου, screening, ώστε να μην επιστρέφουν αυτοί που δεν πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες τους. Με αυτήν την ε, παρατήρηση σας ευχαριστώ και πάλι που μας προσκαλέσατε και είμαι στη διάθεσή σας αν έχετε ερωτήσεις προς εμάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σάκρε. Ίσως να υπάρχουν αργότερα ερωτήσεις. Πάντως σας ευχαριστούμε. Και τώρα μια σύντομη ενημέρωση από την ε, ομάδα δράσης του ΟΗΕ, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης, που επισκέφθηκε την Λιβύη το Φεβρουάριο η ομάδα δράσης, η ομάδα κρούσης, ε, σχηματίστηκε από τον Νοέμβριο στην τελευταία σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικανικής Ένωσης για να δούμε τι θα κάνουμε με το θέμα των μεταναστών προσφύγων και αυτού τον άσυλο που ακολουθούν ε, δυσχερείς οδούς διέλευσης. Έχουμε ήδη συζητήσει με την ύπατη αρμοστία. Έχουμε τον κύριο Μορντή λοιπόν και τον κύριο Πικέ. Ε, ο ένας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο άλλος από την ΕΕΔ. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Ο κύριος Μορντή πρώτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σάιμον. Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Ένα σημείο μόνο για τα πρακτικά για να επισημάνω ότι υπάρχουν διάφορα σχέδια και δραστηριότητες όπως αυτό που αφού από την Επατή Αρμοστία, χρηματοδοτούμενα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι σημαντικό αυτό να το υπογραμμίσουμε γιατί έχουμε να κάνουμε μια δύσκολη κατάσταση με δύσκολο εταίρο και ίσως μερικές φορέ. Δίδεται η εντύπωση ότι έχει περισσότερο κατασταλτική προσέγγιση η Ευρωπαϊκή Ένωση και λιγότερο προσέγγιση προστασίας. Και έτσι αυτά που κάνουμε σε συνεργασία και με την υπατή αρμοστία πολλές φορές παραγνωρίζονται. Ε, για την αποστολή λοιπόν στις 21 και 22 του Φεβρουαρίου καταφέραμε να επισκεφθούμε και την, την και την Τρίπολη μαζί με τον Επιτροπό για τα Κοινωνικά Δικαιώματα της Αφρικανικής Ένωσης και συναδέλφους από την Υπατή Αρμοστία και από την Διεθνή Οργανώση Μετανάστευσης και τον συνάδελφο Κούρσεν Μπλέφοφ και τον κύριο Ποπόφσκι, αντίστοιχα από την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, και τη Γενική Διεύθυνση μετανάστευση. Ήταν ε, ενδιαφέρουσα αυτή η επίσκεψη. Είχαμε καιρό να μεταβούμε στη Λιβύη. Μα επέτρεψε να παρακολουθήσουμε συζητήσει και να συνεχίσουμε συζητήσει που είχαν γίνει ήδη στην Αμπιτζάν, στην Σύνοδο Ευρωπαϊκής, Ευρωπαϊκή Ένωση με τι χώρε Αφρική. Μπορώ να σα δώσω λοιπόν κάποιε εξελίξεις ε, σε σχέση και τι δικές μας θέσεις. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ε, συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον Πρόεδρο της ομάδας ε, της προστασίας των συνόρων, επικεφαλής της ακτοφυλακής, από τον εκπρόσωπο της, των κέντρων κράτησης για αυτούς που ε, θεωρούνται από τις λιβικές αρχές ε, παράνομοι μετανάστες. Πήγαμε στο κέντρο Ταρίκα κοντά στην, ε, Λιβύη, κοντά στην Τρίπολη της Λιβύης και νομίζω ότι είδαμε και προσήλωση στις πολιτικές λύσεις αλλά και προσέγγιση για το μέλλον, λύσεις που μπορέσαμε να εξετάσουμε από πρώτο χέρι και γιατί το κέντρο αυτό, όντα κοντά στην Τρίπολη, είναι το καλύτερο, φανταζόμαστε. Οπωσδήποτε δίνει και μια εικόνα των δυσκολιών που έχουν όλα αυτά τα κέντρα υποδοχή να αντιμετωπίσουν. Ε, μια γενική τοποθέτηση, καταρχά. Αν δούμε τους ε, δρόμους ε, που διασχίζουν την κεντρική Μεσόγειο και όλους αυτούς που φτάνουν στην Ιταλία από την Αφρική. Έχουμε μειωσεί κατά 66% των αφήξεων σε σχέση με τις 5 Μαρτίου του 2017 μέσα σε ένα χρόνο. Επομένως είχαμε μόλις 5.000 αφήξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2018 μέχρι τώρα. Κάποια στοιχεία επίσης ενδιαφέρονται είναι τα εξής, ότι αν κοιτάξει κανείς ποιες είναι οι χώρες αναχώρησης προελεύσεως, έχουμε μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 3.700 που αφικνούνται στην Ιταλία από τη Λιβύη, Επομένως, η συντριπτική πλειοψηφία των, ε, των αφικνουμένων στην Ιταλία είναι Λίβοι. Ωστόσο, έχουμε και σημαντική αύξηση από τους ε, αφικνουμένους από την, την Ισία, 1100 περίπου, δεύτερη θέση με αρκετά μεγάλη διαφορά. Ε, τα στοιχεία αντίστοιχα με αυτά που είχαμε πέρσι. Οι εθνικότητε τώρα από αυτόν περνούν από τη Λιβύη την Τινησία. Έχουμε ισχυρή παρουσία των Ερυθρέων, ένα τέταρτο των συνολικών αφήξεων στην Ιταλία για το 2018. Δεύτερη όμως πλέον αναδεικνύεται η την Ισία με ένα πέμπτο των αφήξεων και ενδιαφέρον είναι ότι για πρώτη φορά διαπιστώνουμε αφήξεις Λιβύων πολιτών. Κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν είχε καταγραφεί σε σημαντικά τουλάχιστον ποσοστά για το 2018. για τη δουλειά και τις συζητήσεις μας στην επίσκεψη αυτή. Οι συνάδελφοι από την είπα ότι αρμοστοί επεσήμαναν κάποια ζητήματα. Ένα από αυτά είναι που ε, πάλι με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση φέρνει αποτελέσματα είναι η εκένωση προσφύγων από τη Λιβύη 1334 και πάλι στο Παρίσι σήμερα με τις συζητήσεις που συνεχίζουν τις ε, προσπάθειες αυτές σημειώνεται ότι υπάρχει βούληση και διάθεση για περαιτέρω με την κατάσταση αλλά και επιτάχυνση της ε, ε, επεξεργασίας των ατομικών ε, αιτήσεων. Επομένως ε, και δεδομένου ότι έχουμε αρκετές δεσμεύσεις από τα κράτη-μέλη για την υλοποίηση των προϋποθέσεων μετεγκατάστασης που ξέρετε ότι έχουμε συζητήσει από τις δεσμεύσεις που ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο για 50.000 ε, επανα επανεγκαταστάσεις, μετεγκαταστάσεις. Έχουμε υλοποίηση των 40.000 από αυτές. Κάποια μεγάλα κράτη ακόμη πρέπει να αναλάβουν τη δέσμευση και 7.000 καλύπτουν τα προφίλ της Κεντρικής ε, Μεσογείου, αλλά και προελεύσεις από τον Ήγηρα και άλλες χώρες. Περίπου 3.500 ε, δεσμεύσεις αφορούν τέτοιες προελεύσεις. Άρα βελτιώνεται η κατάσταση, αλλά χρειάζεται ακόμη περισσότερη προσπάθεια και από τα κράτη-μέλη και από την υπατιαρμοστία, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων, γιατί δεν θέλουμε να θεωρηθεί να θεωρήσει ο Νίγηρας ότι έχει παγιδευτεί και ότι δεν βρίσκει λύση. Πρέπει να δώσουμε μια μόνιμη λύση και πρέπει ε, να δείξουν όλη την ίδια κατανόηση. Επίσης σημαντικό είναι και το έχουμε αναλάβει μαζί με την Οργάνωση για τη Μετανάστευση, Διεθνή Οργάνωση Μετανάστευσης και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, για πάνω από 7.000 επαναπατρισμούς, ασφαλείς επαναπατρισμούς από τη Λιβύη κατά τη διάρκεια του 2017 και πιστεύω ότι μπορούμε σύντομα να έχουμε καλύψει τα ποσοστά των 15.000 επαναπατρισμών, ε, τη δέσμευση δηλαδή του, ε, της Αμπιτζάν μέχρι το Νοέμβριο. Πολλά ακόμα μένουν να γίνουν βεβαίως αν δούμε τα κέντρα κράτησης. Ένα από τα... Μία από τις δεσπιστώσεις είναι ότι μειώνονται τα νούμερα. Βεβαίως δεν είναι καθόλου ακριβής η επιστήμη κατά μέτρηση. Αυτή πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός όταν ε, δίνει στατιστικά στοιχεία γιατί υπάρχουν κέντρα κράτησης που δεν ελέγχει η κεντρική κυβέρνηση της Λιβύης. Ωστόσο ε, πάλι αυτά είναι τα στατιστικά που χρησιμοποιεί και η Διεθνής Οργάνωση Μετανάστευσης. Στο Σεπτέμβριο του 2017 είχαμε 22.000 μετανάστες στα κέντρα κράτησης υπό τον έλεγχο της ε, Διεθνούς Οργάνωσης για τη Μετανάστευση τώρα έχουν πέσει στο 1 τρίτο και νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι και οι Λίβοι, οι ε, Λιβικές αρχές με τις οποίες συνεργαζόμαστε προσπαθούν να εξασφαλίσουν την ε, ριζική μείωση του αριθμού των κρατουμένων στα κέντρα κράτησης. Έτσι λοιπόν απευθύνουμε έκκληση στους συναδέλφους της ΥΠΑ της Αρμοστίας έτσι ότι ώστε η δέσμευση για την ε, αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών, ε, των ε, αλλοδαπών που βρίσκονται στα κέντρα κράτησης, να προχωρήσει ταχύτερα. Και βέβαια και η θεωρήση θεωτηρίου για έξοδο από τη Λιβύη είναι απαραίτητο να προχωρούν ταχύτερα. Είναι αυτό μεγάλο πρόσκομο ώστε να μπορούν είτε να επαναπατριστούν είτε να περάσουν στον Νίγηρα. Ενδιαφέρον επίση είναι το γεγονό ότι την προηγούμενη εβδομάδα η DCIM, η ηγεσία τη καλύτερα, μα έδωσε ένα μήνυμα ότι θα περίμενε να κλείσουν, δει ένα μήνυμα ότι θα κλείσουν τα κέντρα κράτηση. Ε, μπορούμε να περιμένουμε την υλοποίηση αυτή τη δέσμευσης, βεβαίω, όχι αμέσω, αλλά τα κέντρα χρειάζονται και ανακαίνιση και εξυγχρονισμό. Δεν είναι καλέ συνθήκε κράτηση αυτή τη στιγμή. Ε, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου πήρα κάποιες φωτογραφίες και πρέπει να σας πω ότι και ότι αυτή ήταν η πιο επιτυχημένη περίπτωση κέντρου κράτους. Ε, εγώ ή, οσδήποτε από την οικογένειά μου δεν φαντάζομαι να μπορούσαμε να αντέξουμε να μείνουμε σε ένα τέτοιο κέντρο κράτησης, αλλά πρέπει να πιέσουμε προς, προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης πρέπει να συνεχιστεί η δουλειά για τη δημιουργία ενός συνολικού και, και ανιχνεύσιμου θα έλεγα συστήματος ε, καταγραφής των μεταναστών. Η εκτοφυλακή της Λιβύης αυτή τη στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους συγκεκριμένα έχει διασώσει 31.000 ε, ανθρώπους, γι' αυτό βλέπουμε και σημαντική μείωση ε, της απώλειας ανθρώπινης ζωής ε, στα νερά της Μεσογείου. Ωστόσο πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί που διασώζονται από την ακτοφυλακή της Λιβύης, που εκφορτώνονται και ε, στη συνέχεια που πηγαίνουν, που μεταβαίνουν. Υπάρχει ένα σύστημα λοιπόν με την υπατή αρμοστία και την ε, διεθνή υπηρεσία, ε, το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση, για να καταγράψουμε τα νούμερα αυτά και γι' αυτό θα πρέπει να πιέσουμε περισσότερο τι κυβερνήσει να μα δώσουν στοιχεία. Κάποιο άνοιγμα βλέπουμε, κάποια καλή διάθεση δηλαδή βλέπουμε. Βεβαίω θα χρειαστεί να τυποποιηθούν οι διαδικασίε έτσι ώστε να καταγράφεται επακριβώ ε, ποιο αναλαμβάνει τι, ποια διαδικασία λειτουργεί, πώ γίνεται η εκφόρτωση, και επίσης πρέπει η ταχύτερη υιοθέτηση αυτών των κοινών διαδικασιών να μας βοηθήσει σε μια πλήρη καταγραφή στοιχείων, σε ένα σύστημα δηλαδή ε, που θα μπορούν να καταγράφονται και να αναγνωρίζονται οι ε, ενδιαφερομένοι μετανάστες. Πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα για πιο περιορισμένο χρόνο αυθαίρετης κράτησης, έτσι ώστε να περάσουμε από ένα σύστημα κράτησης, σταδιακά βέβαια, σε ένα σύστημα υποδοχής. Και άμεσα αποτέλεσμα της αποστολής και θετικό πρέπει να επισημανώ καταλήγοντας, είναι ότι οι αρχές της Λιβύης παρέδωσαν επέδωσα μόνο στις αρχές της ΥΠΑ της Αρμοστίας ε, επιστολή που τους επιτρέπει να ε, επισκεφθούν τις διάφορες εγκαταστάσεις. Αυτό είναι μια σημαντική πρόοδος και επίσης είναι πολύ σημαντικό να ικανοποιηθεί η ανάγκη για προστασία των παιδιών και των ευάλωτων ε, ατόμων. Βέβαια μέχρι να συμβεί αυτό θα πρέπει να εκδηλώσουμε βούληση να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και να εργαστούμε καταπώνητα ώστε να στηρίξουμε αυτού οι οποίοι βρίσκονται παγιδευμένοι στα κέντρα κράτη. Μέχρι ότου αναπτυχθούν όλε αυτέ οι εναλλακτικέ. Τελευταία παρατήρηση, τελευταίο σημείο που θέλω να επισημάνω είναι η συζήτηση που είχαμε για το είδο υποστήριξη που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε σε δημοτικές αρχές αυτή την εβδομάδα. Και αν δεν απατώμε στις 7 Μαρτίου έχουμε μία συζήτηση για τα θέματα ακριβώς της Αφρικής που θα δώσει τη χρηματοδότηση των 50 εκατομμυρίων για το ευρωπαϊκό καταπίστευμα στη ε, διαχείριση της Ιταλικής ε, Αρχής και των Ευρωπαϊκών αντίστοιχα για να υποστηριχθούν οι δημοτικές αρχές που χρησιμοποιούν ε, τη Λιβύη και μετά την Μεσόγειο να περάσουν στην Ιταλία. Άλλο ένα σημείο που θέλω να επισημάνω για την ακτοφυλακή της Λιβύης και επίσης ένα από τα σημεία που έχουμε με έμφαση υπογραμμίσει στη συζήτηση με τους εταίρους μας πέραν της εκφόρτωσης ε, έχουμε να κάνουμε με την αποτελεσματική παρακολούθηση που προχωρά αυτή τη στιγμή. Θα έχετε δει φαντάζομαι από τις ενημερώσεις από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης του θα θέλει να πει κάτι. Έχουμε επιλέξει τρεις δρόμους βελτίωσης της δουλειάς. Καταρχάς συλλογή πληροφοριών. Δεύτερον εξ αποστάσεως ε, παρακολούθηση στη θάλασσα, στα διεθνή ύδατα και τρίτον περιοδικές ε, συναντήσεις έτσι ώστε να ενημερωνόμαστε από τις λιβικές αρχές, την ε, ακτοφυλακή και το προσωπικό της επιχείρησης Σοφία γιατί έτσι μπορούμε να δώσουμε και στο προσωπικό και στους Λιβύους εταίρους ενημέρωση, κατάρτιση πάνω στη δουλειά αυτή, η πρακτική κατάρτιση δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα αυτό στηρίζει και την υπατή αρμοστία, η οποία με δική μας ε, χρηματοδότηση υπογραμμίζω έχει προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση σε Λιβύους αξιωματούχους και αυτό ταυτόχρονα νομίζω δείχνει ότι και το προσωπικό ή αξιωματούχοι οι οποίοι χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια κάνουν πολύ καλύτερα τη δουλειά τους. Mm. Θα σταματήσω εδώ, πολλά ακόμα θα μπορούσα να πω ασφαλώς, αλλά νομίζω ότι ήταν μια καλή επικοδομητική επίσκεψη με ε, καλό και χρήσιμο διάλογο και ταυτόχρονα αποτελεί την απαρχή μιας διαδικασίας που ελπίζουμε ότι θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε περισσότερο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε και τώρα από την εξωτερική μπλήση εξωτερική δράση τέλο πάντων, κύριο Πικέ. Θα γυρίσω το λόγο για 5-10 λεπτά και θα ακολουθήσουν ερωτήσει από του βουλευτέ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία και κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομο γιατί σα τα είπε πάρα πολύ αναλυτικά ο κύριο. Ε, Διευθυντής όσον αφορά την κοινή επίσκεψη στην Τριπολίτιδα. Από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Περισσεξιτικής Δράσης, ε, ε, ΟΗΕ και είχαμε τη συνάντηση της Άντης και αυτή τη συνάντηση κορυφής και την Task Force όσον αφορά τα θέματα μετανάστευσης. Εκεί έλαβαν μέρος και οι τρεις πλευρές. Οπότε και είπαμε ότι αποτελεί ευκαιρία απαρχής για νέα συνεργασία, ούτω ώστε να έχουμε παγίωση της νόμης μετανάστευση στην ε, Λιβύη. Αυτό το πετύχουμε με πολλούς τρόπους. Πρώτα-πρώτα, χάρη στη συνάντηση κορυφής, η εμπλοκή της χώρας τώρα είναι πιο ρεαλιστική, πιο δυναμική, κάτω με τον επαφών μαζί μας και όσον αφορά την πολιτική που ακολουθεί και επίσης έχουμε τώρα πιο στενή συνεργασία και υποστήριξη από πλευράς των Αφρικανικών χωρών. Η, της δηλαδή προέλευσης των ε, παρανομών μεταναστών στην Λιβύη. Επομένως, κατά πολλούς τρόπους, βοήθησε συνάντηση κορυφής και επίσης η Task Force. Όσον αφορά τώρα από πλευρά των Λιβικών αρχών, η ομάδα εργασία για την μετανάστευση που σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης ε, η Λιβύη έχει συγκροτήσει και διατηρήσε λειτουργία ασχολήθηκε με το θέμα του να υπάρχει μια ουσιαστική πλατφόρμα για διάλογο, για καθορισμό προτεραιοτήτων στο μέλλον. Τι σημαίνει αυτό, πέραν από όσων όσον σας είπε ο κύριος Μόρτιο. Από πλευρά τη υπηρεσία τη έχουμε προσθέσουμε τα εξή. Πρώτα-πρώτα, Η αποστολή βοήθειας διαχείρισης των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Λιβύη έχει ξεκινήσει. Έχει εγκατασταθεί η αποστολή στην α, ε, ε, Λιβύη από τον Δεκέμβριο, είναι πλήρως λειτουργική. Οπότε τώρα η αρρωγή μας προς την χώρα είναι πιο ουσιαστική. Συνεργαζόμαστε με τις αρχές της χώρας, Υπουργείο Δικαιοσύνη, Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά ακτοφυλακή, ε, συνοριοφυλακή της χώρας και είχαμε εκένωση προς ε, την Τίνιδα Πάντως έγινε την παρουσία μας στην Τριπολίτη και θα πάει την προσωπία μας εάν επιτρέπει η κατάσταση ασφαλείας. Αυτό θα γίνεται μία με δύο φορές την εβδομάδα. Η επιχείρηση Σοφία συνεχίζει να διασώζει μετανάστες, συνεχίζεται αυτό το επικίνδυνο ταξίδι προς τις νότιες ακτές της Ευρώπης και συνεχίζεται η εκπαίδευση της ε, λιβικής ακτοφυλακής. Εκπαίδευση όχι μόνο όσον αφορά τη διαχείριση της ε, λάθρομετανάστευσης κατά θάλασσα, αλλά και όσον αφορά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε συνεργασία με την ε, υπηρεσία της υπάτης εκπροσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ανανεώνεται η εντολή της Σοφία για να καλυφθεί η υπόθεση μετανάστευση. Τέλος, θα πρέπει να συνεχίσουμε να λοιπόν υπόψη μας ότι η συνεργασία με την χώρα συνεχίζει να διέπεται από κάποιους περιορισμούς, από την αστάθεια στην χώρα, από την διακυβέρνηση που διακρίνεται από αστάθεια και από την έλλειψη συνθήκων ασφαλείας. Έχουμε πετύχει σε αυτό το μέτωπο κάποιες βελτιώσεις, αλλά η δυσάρεστη κατάσταση για τις συνθήκες ασφαλείας είναι πάρα πολύ ευμετάβλητη, και πότε προκύπτουν συνέπειες πρακτικές όσον αφορά την υπόθεση της συνεργασίας μας. Εμείς πάντως θα πρέπει να συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τον ΟΗΕ για να υπάρξει κάποια βιώσιμη διαρκής λύση με τη διακυβέρνηση της χώρας ούτως ώστε να Έχουμε εκλογές μόλις ε, αυτό καταστεί δυνατόν. Έχουμε κάποιο είδους ε, ενοποίηση των στατικών παραστατικών ομάδων υπό πολιτική ενιαία διοίκηση. Πώς ξέρετε αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, πολύ σημαντικό. για ε, κάποιος θέλει να έχει συνθήκες κράτους δικαίου στη χώρα. Οπότε θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την μετανάστευση, αυτά τα οποία έθιξε ο κύριος Μόρτζιο. τους νέους διαδρόμους, τις νέες διαδρομές με τις νέες της χώρας προσπαθούμε να φροντίσουμε και να δούμε τι θα γίνει με την περιφερειακή διάσταση μια που θέλουμε να συνεχιστεί ο διάλογος και η συνεργασία με τους γείτονες της χώρας προς Νότο, Ανατολή και Δύση και ευρύτερα στις χώρες νοτίου της ε, Σαχάρας. Οπότε και να ασχοληθούμε με τις απότερες, τις βασικότερες αιτίες της μετανάστευσης. Ευχαριστώ. Και τώρα έρθει η ώρα των ε, συναδέλφων. Παρακαλώ να δύο ο καθένας. Κύριο Στέτη είναι πρώτος, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει κύριο Στέτινα. Παρακαλώ, φορέστε τα ακουστικά σας και θα σας τα πω στα τσεχικά. Πρώτα πρώτα, να ευχαριστήσουμε την κυρία Σάχλου για τα όσα μας παρουσίασε, για όλη αυτή την ενημέρωση. όμως και ο διηγητής του Λαϊκού Κόμματος για την έκθεση που έχει ετοιμάσει η Επιτροπή μας διατυπώνουμε και κάποιες συστάσεις προς το Συμβούλιο και την υπατή εκπρόσωπο. Όσα ήδη έχετε κάνει αξίζουν του επένου μας. Και στο κείμενο ακριβώ αναφέρουμε και σε τροπολογίες ο, τα θέματα της προσπάθειάς σας για την ε, εκένωση. Είπαμε ότι περίπου 5.000 σήμερα ακόμη βρίσκονται σε αυτά τα κέντρα κράτησης που ελεγχόνται από την κυβέρνηση. Μπορείτε να μας δώσετε μια ιδέα για το πόσοι σήμερα κρατούνται σε κάποια κέντρα που δεν είναι υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης. Δεύτερη ερώτηση. Μπορείτε να μας πείτε ποιες από τις δραστηριότητες στη Λιβύη χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Επίσης, Επαναλαμβάνω, πόσοι βρίσκονται σε κάποια κέντρα κράτηση τα οποία δεν έρχονται από την κυβέρνηση. Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε το ποια είναι η συμμετοχή των Ευρωπαϊκών Ταμείων στις δραστηριότητε αυτές. Σας ευχαριστώ. Έχω διάφορε ερωτήσεις να σας υποβάλω. Ευχαριστούμε που ήρθατε και ευχαριστούμε την εκπρόσωπο τη ΥΠΑ της Αρμαστίας λέει η κυρία Μπιόρ, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι το έργο σας και σας ε, ερωτώ. Όσον αφορά τις εθελοντικές ε, επιστροφές, επαναπατρισμούς τέλο πάντων που οργανώνεται, ε, υπάρχει ο κίνδυνος επαναπροώθησης πολλών εξ αυτών. Δεν μπορεί να έχετε πρόσβαση σε όλους αυτούς. Άρα πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνει αυτή η επαναπρόθεση. Επίση. τι γίνεται για το ότι έχετε πρόσβαση σε περιορισμένο αριθμό εθνικοτήτων. Πώς να βελτιωθεί η κατάσταση σε αυτό το μέτωπο. Ε, υπάρχει de facto κίνδυνο επαναπρόθεση. Επίση, όσον αφορά τα σημεία απόβαση ή αποβίβασης. Τι γίνεται, πηγαίνει ο, άνθρωπο, ο, κόσμος, ο πηγαίνει από εκεί στα κέντρα κράτηση. Τι μπορεί να γίνει για αυτούς που ζητούν άσυλο. Τι γίνεται με το πρωτόκολλο συνεργασίας ή όπως αλλιώς το λέτε. Θα ήθελα να δω αυτό το πρωτόκολλο συνεργασίας και να ξέρω όσον αφορά αυτά τα σημεία αποβίβασης ποιος έχει ποιες αρμοδιότητες. Έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή το θέμα αυτών των ε, κέντρων και καταβλισμών και δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να χρηματοδοτούμε αυτά τα κέντρα, αυτά τα στρατόπεδα είναι ντροπή. Άρα πώς έχει σημειωθεί πρόοδος και σε αυτό το μέτωπο τέλος όταν όσο αναφέρονται για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Λιβική Εγγραφυλακή είχαμε 50 οι οποίοι πέθαναν οι φωνεύτηκαν ακριβώ λόγω τη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από του Λίβιου. Έχουν ερευνηθεί αυτέ οι υποθέσει. Τι σχεδιάζετε να κάνετε, γιατί έχετε αναφέρει, ξέρω, ότι θέλετε να υπάρχει ένα κέντρο συντονισμού για τη θαλάσσια δραστηριότητα. Δεν υπάρχει κράτο δικαίου. Πώ είναι δυνατόν η Λιβύη να έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για μια συγκεκριμένη ζώνη στη Μεσόγειο. Αυτό είναι ανεύθυνο. Θα ήθελα να με ε, ενημερώσετε πάνω σε αυτό. Αυτά με ανησυχούν και με αυτά μπορώ να μου τα εξηγήσετε. Κυρία Σαρχεντίνη, πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστούμε πάρα πολύ την υπάτη αρμοστία για την προσπάθεια που κάνει και αυτή όσον αφορά το να βγουν οι πρόσφυγες από αυτά τα κέντρα κράτησης αυτούς που πήγατε στον Νίγερ τι ισχύει τους αφήστε εκεί ε, αυτό δεν ήταν λύση να μείνουν εκεί για την υπόλοιπη ζωή τους δεν μπορώ να καταλάβω πως από τη μία πλευρά φροντίζουμε την μετακατάσταση και από την άλλη μεριά εκπαιδεύουμε τους ακτοφύλακες της ε, Λιβύης να σταματήσουν τον κόσμο από το να διασχίσουν την ε, Μεσόγειο. Τους σταματήσουν δηλαδή και να μην τους σώζουν τη ζωή την άλλη μεριά. Δεν θεωρείται, δεν είναι. Ούτε η ούτε η χώρα ασφαλής και ούτε καν τα λιμάνια της χώρας είναι ασφαλή. Δεν νοείται πραγματική συνεργασία με αυτή την χώρα και εκπαιδεύεται τους εκτοφύλακες για το τι θα κάνουν με τους πρόσφυγες εκεί γιατί άμα τους ε, σώσει κάποιο πλοίο που φέρει ευρωπαϊκή σημαία, δεν μπορούμε να μετά να τους αποβιβάζουμε στην ε, Λιβύη. Μα δεν είναι ε, ασφαλείς εκεί οι λιμένες. Αν ήταν ασφαλείς, τους πήγαμε και εμείς να τους αποβιβάσουμε εκεί. Τι γίνεται με τα λιβικά σκάφη. Είναι λάθος Μα πώς ο κόσμος να θέλει να επειδή να διασωθεί τελος πάντων ένα λιβικό σκάφος αφού θα καταλήξει σε μη ασφαλές λιμένα. Ε, γι' αυτό και ξεσπάει βία σε αυτά τα σκάφη. Και μετά την αποβίβαση τι γίνεται, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Το μόνο συμπέρασμα μπορεί να υπάρξει είναι ότι δεν θα έπρεπε σε αυτό το μέτωπο να υπάρξει συνεργασία. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ υποκριτικό εάν δεν κάνουμε κάτι να ξεκαθαριστεί η υπόθεση με την κατάσταση από τον Νίγηρα. Κυρία Βαλέρο, ναι και εγώ μελετώ τη στρατηγική περιορισμού του κινδύνου που έχετε καταθέσει και βλέπω ότι υπογραμμίζεται και το ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων για τα πλοία, για τη διάσωση. και στα πλοία και στη Σαχάρα. Είχα αυτή την Παρασκευή ως μια συνάντηση με μια μη κυβερνητική οργάνωση που ασχολείται με έρευνα και διάσωση και ακόμη τους απασχολεί το γεγονός ότι περιγράφεται ως εγκληματική δραστηριότητά τους και ότι επιπλέον ε, υπάρχει η κατηγορία πως προσελκύουν με τη δραστηριότητά τους ε, τους μετανάστες υποψήφιους να διασχίσουν την ε, Μεσόγειο. Είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει εδώ και πολύ καιρό. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αν έχετε κάτι να σχολιάσετε. Αλλά πάνω απ' όλα για την κατάσταση θέλω να ρωτήσω αν τα πράγματα είναι τόσο άσχημα όσο μας έχουν πει ή εν πάση περιπτώσει τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Και βέβαια για την έρευνα και διάσωση θέλω να απαντήσω στην ερώτησή μου. Ευχαριστώ πολύ Μπόντουλ και ε, μια τελευταία ερώτηση θα δεχθώ. Ξέρω και με συγχωρείτε ότι θα ενοχληθείτε, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ίσως την επόμενη φορά, όχι ότι ε, θα έχουμε κάποιον άλλον την επόμενη φορά, αλλά ίσως την επόμενη φορά η Επιτροπή να μπορεί και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε θέλω να πω. Μπίρκετ, μια τελευταία. Γιατί θέλουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαστε δυνατόν πιο σύντομοι, λέει η κυρία Ζήπηλ. Ε, δεν αμφιβάλλω ότι αυτοί που εμείς ε, έχουμε την τάση να αποκαλούμε λιβική κυβέρνηση ε, κάνουν ό,τι μπορούν. Ωστόσο, αν κοιτάξουμε την καταστροφική κατάσταση και για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, αλλά και για τους ίδιους τους Λιβύους, δεν βλέπω πώς είναι δυνατόν να έχουν πράγματι οργανώσει και επιπλέον, να το οργανώσουν και επιπλέον ε, για το εμπόριο. Πού είναι τα κράτη-μέλη. Πού είναι αυτοί που πρέπει να προσφέρουν την υποστήριξή τους. Δεύτερον, αντιλαμβάνομαι ότι οι μετανάστες που φεύγουν από τα στρατόπεδα αυτά, από τους καταβλισμούς αυτούς, δεν θέλουν να φύγουν με τον κίνδυνο να ξαναβρεθούν στην ίδια κατάσταση. Άρα λοιπόν ίσως θα ήταν μία λύση αυτοί οι άνθρωποι να αποχωρήσουν, να βγουν από τη, από τη Λιβύη. Ωστόσο, και αν καταλαβαίνω καλά είναι περί τους 500.000, μόνο όμως 40.000 είναι διατεθειμένοι να ή έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν άσυλο ή διεθνή προστασία και λυπούμε, αλλά Ντρέπομαι, ντρέπομαι που δεν αναλαμβάνουν σχετικές δεσμεύσεις τα κράτη-μέλη. Ε, έχουμε πάνω από 500 εκατομμύρια πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. 40.000 δεν μπορεί να είναι πρόβλημα για τα κράτη μας. Γι' αυτό λοιπόν ε, το να χρηματοδοτούμε καταβλισμούς και κέντρα κράτηση στη Λιβύη δεν είναι λύση. Θα ήθελα μια ουσιαστική λύση και θα ήθελα και πιο πολλά ε, και από την Υπατή αλλά και από την Επιτροπή, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να μας πούν τι έχει πάει στραβά και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τόσο τώρα μέσω αλλά και με πρόθεσμα. Ευχαριστώ. Βεβαίως πολλά από αυτά που ακούσατε έχουν να κάνουμε μια αποστολή, μια αντιπροσωπεία στη Λιβύη και την, ε, την είδα βεβαίως και παρακαλώ ε, να και εσύ να μας πεις Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σύντομα για μην κατηγορούμε γιατί άκουσα αυτά τα οποία μας ε, είπε η Κνούρ και αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μόρτιου. και ε, βλέπω ότι υπάρχει πέρα μια έλλειψη συγχρονισμού γιατί από τη μια μεριά η Ακνούρ μας λέει ότι χρειάζονται περισσότερο χώρο και χρόνο μάλλον και περιθώρια χρονικά για την ε, μετακίνηση και με την κατάσταση από τον Ήγηρα. Αλλά ο κ. Μόρτζη μας είπε ότι είναι θέμα για κάποιο είδους διαπίστευσης. Ε, και τι να κάνουμε εμείς, πώς να βοηθήσουμε τόσο ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο συντονισμό και συγχρονισμό ενεργειών. Ε, ε, ε εντάξει, όπως είπατε και εσείς με τα λόγω γνώσεων υπάρχει αυτού του είδους η αύξηση των ε, Τινησίων και η κατεύθυνση τους προς ε, την ε, Μεσόγειο. Τι λέτε, ο Πρόεδρος. Είναι βέβαια, θα μπορούσαμε βέβαια να εμβαθύνουμε περισσότερο, αλλά τέλος πάντων ε, έστω έτσι μια φωτογραφική απεικόνιση του τοπίου ας έχουμε. πρώτα πρώτα να μας τα πει πρόσωπος της υπάτης αρμοστίας. λέει η κυρία Σάκρο, να σας πω όσον αφορά ε, για τις ερωτήσεις σας, ότι για αυτούς τους 5.000 που είναι ακόμα, είπατε, σε κάποια κέντρα κράτησης και ποιοι είναι εκτός κυβερνητικού ελέγχου, ε, εμείς, ως μαστία δεν έχουμε την απάντηση εις αυτό. Διότι εμείς δεν έχουμε πρόσβαση, δεν γνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα εκτός κυβερνητικού ελέγχου κέντρα. Το θέμα είναι όταν έχουμε αυτή την ε, κατάσταση εκτά των ανάγκη, έχουμε μετανάστες και πρόσφυγες εδώ σαν Σαμπράτα και ξέρουμε ότι κάπου είναι. Οπότε ο IOM και εμείς ε, έχουμε πρόσβαση στα επίσημα κέντρα ε, υποδοχής, κράτησης, τέλος πάντων. Ναι, υπάρχουν κέντρα εκτός του ελέγχου πόσα είναι, που είναι, δεν γνωρίζουμε. Όταν μάθουμε θα επικοινωνήσουμε άμεσα με την κυβέρνηση να μεταβούμε εκεί και να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία που έχουμε τώρα όσον αφορά τις δραστηριότητε που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ένωση χρηματοδοτεί σχεδόν το σύνολο των δραστηριοτήτων και επεμβάσεων μας στη χώρα. Τώρα για τον μηχανισμό ε, της ε, και Ένωσης και αυτό την κατάρτιση, μεταφορά κλπ. Δεν καλύπτονται όλες οι επεμβάσεις, αλλά συμμετέχει στην πρικοδότηση όλων αυτών των ε, δρασιών. Έχουμε αυτά τα 13 εκατομμύρια για την Αφρική που πάνε όλα στη Λιβύη και θα έχουμε άλλα 5-6 μας έχουν υποσχεθεί 5-6 ευρώ. Αυτά θα προωθούν από την ΕΚΟ και από τα καταπιστεύματα. Επίσης, είναι σημαντικό να αναδείξουμε το ότι για αυτό το, το, το, το κέντρο Transit, της εκτάκτων ανάγκης που ενέκριναν οι ελληνικές αρχές ε, και αυτό πρόκειται να επανενεργοποιηθεί χάρη στα κοινοτικά κονδύλια τώρα όσον αφορά το ότι έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες εθνικότητες και όσον αφορά τα όρια και τους περιορισμούς μας για την επαναπρόθεση, ε, όταν μας ζητήσανε να πάμε στη χώρα και να ασχοληθούμε περισσότερο μετά τη Σομαλία ε, την κρίση που σοβούσε ε, δεκαετία του 90, η, η χώρα ε, δεν είναι τόσο κατανόηση στα θέματα του ασύλου. Και οι πρόσφυγες πάντοτε θέλουν να ενταχθούν στην τοπική κοινωνία. Ε, αυτό το θέλει η κυβέρνηση τη χώρα. Ε, γι' αυτό λοιπόν και παραδοσιακά δουλεύουμε με συγκεκριμένες ε, εθνικότητε του οποίους μετεγκαθιστούμε. Και Έχουμε τους παραδοσιακούς Άραβες, ε, γιατί αυτοί πιο εύκολα μπορούν να πάνε στη χώρα. Θεωρούνται αδελφοί, Παρελιστίνοι, Ιρακινοί, Σύριοι και για τους ε, Αφρικανούς. Είχαμε συμφωνήσει με τους Λίβιους ότι θα τους βρούμε λύση εκτός της χώρας. Οπότε και η διεθνής κοινότητα Προσπαθεί να δει τι θα γίνει με τις λοιπές εθνικότητες τώρα για την αποβίβαση και τι γίνεται με τους αποβιβαζόμενους. Έχουμε είπαμε 12 τέτοια σημεία αποβίβασης. Συντονισμός γίνεται με τον IOM. Πάνε στα τόπεδα κράτη, ο κόσμος, καταγράφονται εκεί. Εξετάζεται ο βαθμός ε, του πόσο ευάλωτη είναι τέλος πάντων και μετά πάνω στο CDC τα κέντρα φιλοξενίας που βρίσκονται υπό την αιγίδα της ΥΠΑ της Αρμοστίας, οπότε γίνεται εκεί η ταυτοποίηση και μπαίνουν σε κάποιες λίστες για την ΕΕ Ένωση. Τώρα, τελευταία ερώτηση που εμεί θα μπορούσαμε να απαντήσουμε, υπάρχει θέμα χρόνου, ποια κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί για την υπόθεση με την κατάσταση από τον Νίγηρα. Η Γαλλία ήδη έχει συμμετάσχει δύο-τρεις αποστολές, η Ελβετία και άλλες χώρες που έχουν δεσμευτεί σχετικώς. Ιταλία, Νορβηγία, Σουηδία και Μάλτα, αλλά και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι πώς θα γίνουν οι συνέντευξες, πώς θα γίνουν οι έλεγχοι ασφαλείας. Ε, με αυτό παίρνει πολύ χρόνο. Που τώρα έχουμε 25 πρόσωπα που πηγαίνουν από Νίγηρα προς Γαλλία. Πάνε ή πήγαν τέλο πάντων. Μόνο, μόνο 25. Ευχαριστούμε πολύ και με συγχωρείτε κυρία Γιουροβά για την καθυστέρηση. Ήταν ευαίσθητο το θέμα και σημαντικό να ακούσουμε τις απαντήσεις στις συγκεκριμένε ερωτήσεις των ε, βουλευτών. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μορντή και τον κύριο Πικέ γιατί μας ε, εξέθεσαν μέσα στον πολύτιμο χρόνο τους όλα αυτά τα στοιχεία και θα ήταν ε, καλό να δοθεί και συνέχεια στις βασικές παρατηρήσεις των ε, βουλευτών. Ναι, πολύ, πολύ σύντομα. Οι ακριβείς αριθμοί δεν είναι και θετική επιστήμη αυτή. Απλώς ε, ο Οργανισμός Ασύλου και Μετανάστευσης δημοσίευσε αριθμούς τον περασμένο μηνό μιλάμε για 750.000 μετανάστες συνολικά στη Λιβύη αυτή τη στιγμή, αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις, γιατί άλλαξε η μεθοδολογία της καταγραφής. Και δεν θα συμφωνήσω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικοί θέλουν απλώς να ταξιδέψουν και να ε, εργαστούν στη Λιβύη και βρίσκονται σε δυσχερεί συνθήκες. Για τις υποσχέσεις περί με την κατάσταση και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε 40.000 θέσεις αυτή τη στιγμή και για την Ανατολική Μεσόγειο και για την ε, Κεντρική Μεσόγειο. Αν δούμε την Κεντρική Μεσόγειο, νομίζω 14 Ιθαγένειες καλύπτονται 7.000 θέσεις έχουν υποσχεθεί τα κράτη-μέλη και από αυτές συγκεκριμένα 3.425 ε, θα υποστηρίξουν όσα κάνει αυτή τη στιγμή η πατιαρμοστία με τον μηχανισμό άμεσης ε, ε, διαμετακόμιση. Έχουμε από την Ιταλία, την Ελβετία και την Γαλλία θέσεις που έχουν δεσμευτεί. Και έχουμε επίσης 1.300 ακόμη που Περιμένουμε σύντομα να αποσαφινιστούν. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλύψει τον αριθμό των ανθρώπων που έχει η πατερμοστία στον Ήγηρα και θα μπορέσει να τα καλύψει στο άμεσο μέλλον. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Αυτή τη στιγμή, καθώ μιλάμε, υπάρχει συνάντηση αυτού που λέγεται τη βασική ομάδα βασική ομάδα ε, για την ε, μετεγκατάσταση από τη Μεσόγειο ε, και γίνεται στο Παρίσι με προεδρία της Γαλλίας, ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να επιταχυνθεί με την κατάσταση, ή ε, με την κατάσταση από τον Ήγηρα, αρκεί να υπάρξει συντονισμός των Υπουργείων Εσωτερικών στο Μιάν στις 16 Μαρτίου, νομίζω. Και είναι σημαντική και η έκκληση τη ΥΠΑ Αρμοστία για τη χρηματοδότηση, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να έχει μια σφαιρική προσέγγιση. Την περασμένη εβδομάδα, μόλι, για να σα δώσω ένα παράδειγμα, υιοθετήσαμε ένα παράδειγμα αξία 150 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ των διαφορετικών ε, παραθύρων που προσφέρει, θηριδών που προσφέρει το καταπίστευμα για την προστασία προσφύγων και μεταναστών και τα κονδύλια αυτά θα αναλάβουν να τα εκτελέσουν η ε, ε, τη αρμοστία και ο Οργανισμό Ασύλου. Τώρα για την ακτοφυλακή και γιατί επιμένουν στην εκπαίδευσή του. Διότι πολλά ατυχήματα έχουν ε, επισυμβεί σε φάση που τα σκάφη βρισκόταν στα χωρικά έδατα τη Λιβύη. Δεν είχαν σκάφη για να κάνουν, κάνουν επιχειρήσεις διάσωσης ε, οι ακτοφυλακές ε, πέρσι, πριν 1,5 χρόνο. Παιδεύσαμε 251 ακτοφύλακε στην Ιταλία και με πολύ ισχυρό μηχανισμό ελέγχου, ώστε όσοι έχουν ερωτηματικά να ξέρουν ότι δεν θα υποφεληθούν όσοι δεν πρέπει από την ε, εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έπειτα η ΕΕΔ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχουν το κατά πόσον αυτά λειτουργούν. Πάντως δεν υπάρχει επιβολία. Ε, διασώζονται ζωές και κάποιοι έχουν ε, ε, διασωθεί από σκάφη τα οποία ιδάλω μπορεί να του είχαν χτυπήσει και να είχαν χάσει τη ζωή του. Εδώ για τα κέντρα κράτηση. Βεβαίω ε, η πολιτική μα είναι να χρησιμοποιήσουμε χρηματοδότηση και με τον Διεθνή Οργανισμό του Ασύλου να της μετανάστευσης, να φροντίζει να έχουν πρόσβαση και άνθρωποι για να έχουν υγειονομική περίθαλψη, τρόφιμα, νερό, στέγη. Η εναλλακτική ήταν ή αυτό ή τίποτα. Δεν ήταν εύκολη επιλογή, αλλά έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, αυτό που μα αποσχολεί είναι να σωθούν ζωέ. Με πολιτικό βεβαίω στόχο, κάποια στιγμή τα κέντρα να κλείσουν και να γίνουν κέντρα υποδοχή πιο ανοιχτά. Αυτό που θα πρέπει να έχουμε ω πολιτικό στόχο είναι οι άνθρωποι να μην έχουν την ανάγκη να διακινδυνέψουν τη ζωή του ε, μέσα στη Μεσόγειο, εφόσον του προσφέρουμε πραγματική επανεγκατάσταση και να μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους όσοι πραγματικά μπορούν να το κάνουν. Νομίζω ότι εδώ θα ολοκληρώσω. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Διότι θέλει κάποιο να δευτερολογήσει, αλλά και η επιτροπή πρέπει να μπει. Ε, Τζούντιθ, ε, έχουμε έρθει σε δύσκολη θέση τώρα. Η ΕΕΔ πρέπει να μιλήσει και εκείνη δύο λεπτά. Κύριε Πικέ, παρακαλώ. Δύο λεπτά όμω, αν γίνεται, διότι πιεζόμεθα εδώ. Ναι, καταλαβαίνω, Πρόεδρε. Για την χρηματοδότηση των κέντρων υποδοχή, ε, αυτό που είπε και ο κ. Μορντή, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί την λειτουργία των κέντρων κράτηση. Η πω όπω έχει καταστεί σαφή. Θέλει να κλείσουν τα κέντρα αυτά. Και η στήριξη που προσφέρουμε στη Λιβύη είναι μέσω διεθνών οργανισμών με σκοπό να ε, βελτιωθούν οι συνθήκες των όσων κρατούνται στα κέντρα και όχι να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα αυτά όσοι έχουν. Άλλο ερώτημα για το κατά πόσον κοιτάζουμε τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βεβαίως κάνουμε τις σχετικές έρευνες και ανακρίσεις παρά με συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. είπατε εκπρόσωπος έχει απευθυνθεί σε διάφορα μέλη του Κοινοβουλίου, έχει, γράψει, έχει στείλει γραπτή απάντηση στην περίπτωση ενός επεισοδίου με ένα σκάφος ε, από το 2017. Ελπίζω ότι έχετε λάβει την απάντησή της. Νομίζω ότι ήταν ένα σαφές παράδειγμα τον τρόπο που λειτουργούμε σε τέτοιες υποθέσεις. Τέλος, αν τα κάτι μέλη μας υποστηρίζουν, ναι. Παράδειγμα. Η επιχείρηση από την ε, Σόφια, η UNAF, όπου ε, απέδωσαν προσωπικό και σκάφη μου και τα κράτη-μέλη, η, επιχείρηση Ιουμπάμπη, η οποία χρηματοδοτήθηκε κυρίως από τις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών και έπειτα, ιδίως για την Ιταλία, έχει υπάρξει ιδιαίτερα ενεργή για τη σωστή προσέγγιση της διαχείρισης της λαθρομετανάστευσης. Ε, νομίζω ότι από τις ε, απαντήσεις ήταν ε, αναπόφευκτο το να διατυπωθούν και άλλες ερωτήσεις. 30 δευτερόλεπτα κύριε Σαρτζαντίνη παρακαλώ. Πρόεδρε ευχαριστώ. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή επανεγκατάσταση αυτή τη στιγμή. Η Πατιαρμοστία μας λέει ότι υπάρχουν κάποια κράτη και μας δίνει το κατάλογο που έχουν δεσμευθεί. Μετά μας λέει η Επιτροπή ότι 40.000 ε, δεσμεύσεις, δεσμεύσεις 40.000 άτομα, 3.425 αφορούν συγκεκριμένα τον Ήγηρα. Αλλά ούτε η Επιτροπή, ούτε η Πατιαρμοστία κάνουν αυτή τη στιγμή ε, με την κατάσταση. Έτσι λοιπόν, όταν μας το λένε αυτό, κάποιος θα πρέπει να απαντήσει και να πει ε, σε είναι αυτά που μας λέτε. Δεν υπάρχουν τα στοιχεία αυτά. Ας απαντήσει παρακαλώ η Επιτροπή. Η κυρία Γιώραβα ξέρω ότι θα με σφάξει. Είναι σε όρους λίμπε τα 15 λεπτά της υπέρβασης του χρόνου ισοδύναμα με μια ώρα. Δεν ξέρω σε άλλες επιτροπές τι γίνεται, αλλά η Επιτροπή σαν Αν είναι η κυρία Γιώργοβα σύμφωνη, α απαντήσω λοιπόν. Μα όντως γίνεται η μετακατάσταση με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού, 36.000 τα τελευταία δύο χρόνια και συγκεκριμένα, καθώ είπε άλλωστε και ο συναφός από την Υπατή Αρμοστία, 3.500 τους τελευταίους δύο μήνες από τη Λιβύη απευθείας στην Ιταλία επανεγκατάσταση και με 10.000 ε, ευρώ χαρτζηλίκι από τον Ήγερα στη Γαλλία επίσης έχουμε επανεγκατάσταση με χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύο από τη Λιβύα σε κέντρο ε, διαμετακόμισης κατεπίγουσας στη Ρουμανία. Επομένως υπάρχουν αυτές οι επανεγκατάστασεις με τη χρηματοδότηση και η σημερινή συνάντηση του Παρίσι πιστεύω θα διευκολύνει την επιτάχυνση και την αύξηση των αριθμών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Γιάννα Σέντερ ως πρόεδρο Τις αντιπροσωπείας για το μαγκρέπ, ε, θα πάμε, γιατί μπορέσαμε να πάμε στην ε, Λιβύη, θα πάμε ε, πάλι. Επομένως, είναι πολύ καλή συνεργασία με, τις, με την αντιπροσωπεία σας, αλλά και με τις λοιπές υπηρεσίες, Επιτροπή, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Σας ευχαριστώ θερμά λοιπόν και κυρία Γεώροβα, για άλλη μια φορά σας το συγγνώμη για την καθυστέρηση και σας καλώ να έρθετε στην έδρα για να ε, κερδίσουμε χρόνο αγαπητοί συνάδελφοι όσο να αποχωρήσουν ή να αλλάξουν θέση ενδιαφερόμενοι. Ας κάνω εγώ την ε, εισαγωγή για το σημείο 4.3. Σας παρακαλώ μόνο χωρίς φασαρία οι μετακινήσεις. Πρόκειται λοιπόν για διαρθρωμένο διάλογο με την Επίτροπο Βαγιάρη για θέματα καταναλωτών, ισότητας, φύλων και καθώς έρχεται στην έδρα εξηγώ ότι πρόκειται για την υλοποίηση εφαρμογή. Παρακαλώ με ησυχία. Πρόκειται για την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας 2017 και προτεραιοτήτων ε, του 2018. Αυτά θα συζητήσουμε. Περιμένουμε να ακούσουμε από την Επίτροπο. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι που έχουν μείνει στα και εξακολουθούν τι συνομιλίες σας παρακαλώ να δώσετε λίγη προσοχή. Λοιπόν, έχουμε μια σειρά από θέματα να συζητήσουμε. Η κυρία Γιώργο θα μας πει ποιες είναι οι προτεραιότητες του 2018 και πώς έχει προχωρήσει η υλοποίηση του προγράμματος του 2017. Μετά θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων και ερωτήσεων, απαντήσεων ε, και γι' αυτό ζητώντας για άλλη μια φορά συγγνώμη για την καθυστέρηση, δίνω το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να συνεχίσω τον διαρθρωμένο διάλογο μαζί σας. Δεν χρειάζεται να ζητήσετε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ήταν πολύ σημαντικό και σοβαρό το θέμα. Αντιλαμβάνομαι ότι έπρεπε να ολοκληρωθεί η συζήτηση όπως έπρεπε. Ε, τα θέματα μας όμως ε, είδαμε το 2017 ότι πολλά μπορούμε να καταφέρουμε αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία με που έχουν προσφέρει οι, τα μέλη της Επιτροπής σας. Είχαμε πολλά θέματα, ξέρετε, που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Και πρώτον, θα αναφερθώ στα επιτεύγματα του 2017 και τους ε, τρέχοντες τριμερείς διαλόγους. Ε, τα επιτεύγματα του 2017, ε, το γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, PPO, είναι ένα από τα κύρια επιτεύγματα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε όλοι μας τις προσπάθειες ώστε να αναλάβει δράση και λειτουργία το ταχύτερο δυνατό και να ε, πιστούν και τα κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν να ενταχθούν σε αυτή τη διαδικασία. Με ιδιαίτερη χαρά σημειώνω ότι οι κατοχώρε εντάσσονται στο γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα και ελπίζω να ε, αποτελέσει αυτό ενθάρρυνση και για άλλα κράτη. Αυτή τη στιγμή μαζί με τι κατοχώρε 21 κράτη-μέλη συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Φορέα και πρέπει να πω ότι πολύ ενεργητικότητα και χρόνο έχω δαπανίσει για να πείσω και τα άλλα κράτη να ενταχθούν και τα λοιπά κράτη να ενταχθούν στο ε, φορέα αυτό. Επίσης ένα άλλο επιτεύγμα η έκβαση των διαπραγματεύσεων για την ε, αναθεώρηση της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων με πολύ σημαντική και καθοριστική δική σας υποστήριξη. Σας ευχαριστώ θερμά. και πάνω απ' όλα για την παρακολούθηση, τα θέματα του παγώματος εισόδων. για τον κανονισμό 45-2001, για την προστασία των ιδιωτών σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις υπηρεσίες και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια ο κανονισμός Eurojust. Εγώ προσωπικώς ε, έχω ε, στρατευτεί και θα συνεχίσω τις προσπάθειες. Από αύριο κιόλας έχω τριμερή διάλογο για την ολοκλήρωση αυτών των ε, φακέλων. Τώρα για, τον, για την εφαρμογή του, κανονισμού, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων θέλω να σα ενημερώσω. Έχουμε μπροστά μα ένα πολύ σημαντικό ορόσωμο, 25 Μαου συγκεκριμένα, και αναφέρομαι στην θέση σε ισχύ του λεγόμενου GDPR, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Καταγράφουμε την πρόοδο και την ουσιαστική υλοποίηση του κανονισμού και βέβαια την πρόοδο που πρέπει να σημειώσουν και τα κρατημέλη και οι αρχές οι αρμόδιες για την προσέγγιση των προσωπικών δεδομένων και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έτσι ώστε στις 25 Μαΐου να είναι άπαντες έτοιμοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποδεθεί σε προσπάθειες σε συνεργασία με όλους αυτούς τους φορείς για να προχωρήσει αυτό το νομοθέτημα το οποίο θα αλλάξει ριζικά την τωρινή κατάσταση με 28 διαφορετικές ε, ε, και χωριστές αιτήσει με τα όσα προέβλεπε το καθεστώς μέχρι πριν. Τώρα περνούμε στην αρχή της μίας Υπήρου ε, δίνουμε καθοδήγηση ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τους ιδιώτες έτσι ώστε να ε, ε, τους ευαισθητοποιήσουμε, να τους εξηγήσουμε καλύτερα πώς θα ε, λειτουργήσει το νέο σύστημα, το νέο νομοθέτημα μετά τις 25 Μαΐου του 2018. Έχουμε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και για τον πολίτη, ώστε να γνωρίζει τα δικαιώματά του, να μπορεί να τα διεκδικήσει και να τα ασκήσει. Καθολοσορίζουμε την ε, συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σημαντικού εταίρου στην επεξεργασία αυτού του σημαντικού θέματος και για την ευαισθητοποίηση και την παροχή πληροφοριών στα κράτη-μέλη. Ο κανονισμό για την προστασία, γενικό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, GDPR, έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολλέ είναι χώρε που προσπαθούν να τον μιμηθούν. Έχουμε σημαντικέ ε, ε, απόπειρε από χώρε ανά τον κόσμο που ζητούν περισσότερε πληροφορίε. Η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα θεωρούν ότι είναι προτεραιότητά του η υλοποίηση του κανονισμού αυτού. Για την Ιαπωνία συγκεκριμένα έχουμε συμφωνήσει σε έναν οδικό χώρο για, ε, χάρτη συγγνώμη, για την απάλληψη των ε, διαφορών μας ε, με συμπληρωματικούς κανόνες παραδείγματι ώστε να καλυφθούν τα κενά και ιδιαίτερα και συγκεκριμένα το περιεχόμενο και τεχνικές λεπτομέρειες των λύσεων που θα προβληθούν σε σχέση με τους Ιάπωνες εταίρους. Ένα σχέδιο από αυτό στον επόμενο μήνα θα ε, ακολουθηθεί από την ε, συνήθη διαδικασία προσαρμογής. Βεβαίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα, θα εξακολουθεί να ενημερώνεται με τις τεχνικές πληροφορίες που δίνουμε με τη, σε σχέση με την Ιαπωνία αυτό και σε σχέση με την Νότια Κορέα. Θα γίνει η προσαρμογή ε, αναλόγως αλλά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η αναθεώρηση της ε, σχετικής νομοθεσία της Νότια Κορέα. Ελπίζουμε όμω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μέσα στο έτο τι ε, συνομιλίε μα, όπω και η Ιαπωνία και η Κορέα είναι για μα ε, σημαντικό εταίρο, αλλά και σημαντικό παράδειγμα για όλη την περιοχή αυτή στον χώρο τη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Με το πακέτο αυτό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων προσπαθούμε να προσαρμόσουμε του κανόνε στην τεχνολογία, τι τεχνολογικέ εξελίξει, αλλά και στον τομέα βέβαια του ποινικού δικαίου θέλουμε να επεκτείνουμε τι δραστηριότητε αυτέ, Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιστροφή, Επιτροπή θα δημοσιεύσει πρόταση για την διασυνοριακή πρόσβαση σε αρχεία, ηλεκτρονικά αρχεία και αποδεικτικά στοιχεία με κάποια μορφή ε, και αναλόγως της περίπτωσης ε, θα πρόκειται για τρομοκρατία, παιδική πορνογραφία, ε, λαθροδιακίνηση ατόμων, απαγωγές διεθνείς, ζητήματα τα οποία πολύ συχνά απαιτούν για την διαλεύκανσή τους άμεση πρόσβαση στα στοιχεία που δεν επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Υπάρχουν κρατημέλη βέβαια που έχουν καταβάλει προσπάθειες για τη μετώπιση των προβλημάτων αυτόνομα, ωστόσο χρειάζεται μια συνολική και στέρεη προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια προσέγγιση που θα επιτρέψει στις αρμόδιες αρχές να ζητούν από έναν πάροχο υπηρεσιών άλλου κράτους μέλους δεδομένα, λαμβανομένων βεβαίως υπόψη των αρχών της αναλογικότητας και της ε, και το σεβασμού των ε, ασφαλιστικών δικλείδων για την επεξεργασία των στοιχείων και πάντα μέσα στο σεβασμό των θεμελιδών δικαιωμάτων προσβλέπω στη συζήτηση μέσα στις προτάσεις όταν την υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας καλώ να μας υποστηρίξετε ώστε να προχωρήσουμε ταχύτατα σε συμφωνία πριν από τις ευρωεκλογές. Εκ παραλλήλου υπηρεσίες μου και εγώ προσωπικώς παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στις Ηνωμένε Πολιτείε και ιδίως σε σχέση με το πρόσφατο νομοθέτημα Cloud Act το οποίο αναφέρεται στην ε, επεξεργασία δεδομένων ε, πέραν των συνόρων των ΗΠΑ, αλλά και την ομοθεσία τη σχετική με την Google. Εγώ θα επισκεφτώ σε δύο εβδομάδες ε, τις ΗΠΑ. Είμαι αποφασισμένη να συνεργαστώ με τους εταίρους από τις ΗΠΑ προκειμένου να εξασφαλιστεί μια αποτελεσματική χρήση των δεδομένων, αλλά σε σεβασμό του διεθνούς, κειμένου, του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων και ιδιαίτερο θα επιμείνω οι Ηνωμένες να ε, εκπληρώσουν όλες τους τις ε, υποχρεώσεις ε, που απορρέουν από το Privacy Shield και όλες τις συστάσεις που έχουμε διατυπώσει πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει κάποια πρόοδος μετά την αναθεώρηση αυτή, αλλά ακόμη μένουν κάποια βήματα να υλοποιηθούν από πλευράς των Αμερικανικών αρχών. Τα γνωρίζετε καλά. Ο τόνος που, που θα υιοθετήσω συνομιλώντας με τους Αμερικανούς εταίρους θα είναι πολύ σκληρός αυτή τη φορά. Επίσης μια άλλη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει ήδη κατατεθεί, η σύσταση για το παράνομο περιεχόμενο. Η σύσταση που δημοσιεύτηκε μόλι την προηγούμενη εβδομάδα. Πρόκειται για μια σύσταση που ακολουθεί μια συνολική προσέγγιση για κάθε τύπου παράνομο περιεχόμενο. Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητε και εντοπίζοντα λύσεις διαφορετικές όπου αυτό είναι απαραίτητο, καταθέτει μια σειρά και προβάλλει μια σειρά από ε, δικλείδε που εξασφαλίζουν στον πολίτη ε, περιορισμός προ τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσει μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα του, αλλά και τη δυνατότητα για τον πολίτη να ε, απαιτήσει την αφαίρεση περιεχομένου εάν ε, η ανάρτησή του ήταν παράνομη. Και έτσι έχουμε μία ε, ισορροπία καλή σε σχέση με το παράνομο περιεχόμενο και την ανάγκη για την προστασία της ελεύθερης χρήσης του διαδικτύου. Σημαντικό επίσης είναι να υπογραμμίσουμε ότι το κείμενο αντικατοπτρίζει πλήρως το γεγονός ότι τα ε, μέτρα αυτορύθμισης έχουν φέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Έτσι βλέπουμε με τα αποτελέσματα του κώδικα συμπεριφορά σε σχέση με την ε, ρητορική μίσους στο διαδίκτυο. Και θα ήθελα να πω δύο λόγια και για το κράτος δικαίου. Είναι καθοριστική σημασία για τη δουλειά τη Επιτροπή σα. Ξέρω ότι τα έχετε συζητήσει εντελεχώ με τον πρώτο αντιπρόεδρο Τίμερμαν και θα τα συζητήσετε ξανά την επόμενη εβδομάδα. Στο πρόγραμμα εργασιών για το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμπεριλάβει μια νέα πρωτοβουλία για να ενισχύσει την εφαρμογή των κανόνων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναγγελία αυτή τη πρωτοβουλία ε, εντάσσεται στι ε, κοινέ μα προσπάθειε να ενισχύσουμε την εφαρμογή του κράτου δικαίου ώστε να προωθήσουμε και να, κρατήσουμε, να διαφυλάξουμε τι ε, κοινέ ευρωπαϊκέ μα αξίε σε όλα τα κράτη-μέλη. Η πρόταση αυτή έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο και θα αντλήσει διδάγματα από τι εμπειρίε των πρόσφατων ετών. Επίσης θα λάβει επαρκώς υπόψη το έργο του Κοινοβουλίου σχετικά, συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος που υιοθετήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016, το οποίο θα είναι ε, βάση για στοχασμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης, μαζί με το Κοινοβούλιο, θα κοιτάξει να οργανώσει επί Αυστριακής Προεδρίας μία ε, ε, διάσκεψη για τα συστήματα δικαιοσύνης που θα οργανωθεί στο πρώτο τρίμηνο του στο τελευταίο τρίμηνο του 2018. Ε, εν είδη συμπεράσματο, να πω δύο λόγια για την ε, ανάγκη να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην κατάσταση των μειονοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ δεν υπάρχει γενικώ ε, αρμοδιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα πρόσωπα που ανήκουν σε μειονότητε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά τον ε, σεβασμό ή τη συμμόρφωση των κρατών μελών με όλα τα ε, νομοθετήματα που έχουν να κάνουν ε, με την οδηγία για την φιλετική προέλευση, την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Επίσης, συνδράμουμε τα κράτη-μέλη με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ώστε να υπάρχει πλήρης και εντελεχή συμμόρφωση. Για παράδειγμα, η διαδικασία επί παραβάση που εκείνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά διαφόρων κρατών μελών λόγω τη διακριτική μεταχείριση παιδιών Ρωμά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το φθινόπωρο θα υποβάλουμε μία συνολική αξιολόγηση του ευρωπαϊκού πλαισίου και για το πώς έχουν προχωρήσει τα κράτη-μέλη στις εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρωμά. Θα δούμε τις επιδόσεις, τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις, τις δυσκολίες δηλαδή. Ε, εδώ θέλουμε να ενισχύσουμε τους διάφορους, ε, ε, τις διάφορες σκέψεις ε, που μπορεί να υπάρχουν για την κατάρτιση των στρατηγικών για το διάστημα μετά το 2020 και μετά θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε και με την ισότητα των λαών ε, για το δεύτερο τμήμα της στρατηγικής ε, των ΛΟΑΤ που δείχνει ότι οι περισσότερες δράσεις που προτάθηκαν το 2015 έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς αλλά παραμένει η ανάγκη να συγκεντρωθούν δεδομένα. Η διακριτική μεταχείριση βάσης στη σεξουαλικό προσανατολισμό κάποιου ατόμου ή την ταυτότητα του φίλου που μπορεί να έχει είναι κάτι που ε, ακόμη δεν έχει προχωρήσει. Γι' αυτό να ε, θυμίσω ότι σε 15 ομαδικά προγράμματα σε κράτη-μέλη αποδώσαμε χρηματοδότηση. Προγράμματα που προάγουν την ισότητα και την ιδιότητα του πολίτη, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των ακτιβιστών που ασχολούνται με τα θέματα αυτά από τη βάση της κοινωνίας. Ανυπομονώ να ακούσω τι απόψει για τα θέματα αυτά και ό,τι άλλο μπορεί να σα ε, ενδιαφέρει. Ε, σας ευχαριστώ και πάλι για την ε, εξαιρετική σας δουλειά και ε, για την τόσο στενή και αρμονική μας ε, συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των δικαιωμάτων των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, Βέρα, για τη δουλειά σας. Είναι τεράστιο το εύρος του χαρτοφυλακίου σας και έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Πριν πάω στους συντονιστές, να θίξω εγώ κάτι, εφόσον δεν το θίξουν οι συνάδελφοι για το θέμα των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων που θέσατε. Έχουν ήδη αρχίσει να ακούγονται κάποιοι θόρυβοι, να γίνεται θόρυβος από τις ανησυχίες που έχουν υψωθεί. Λόγω χάρη ποια θα είναι η προθεσμία, αν υπάρχει κάποια αναβολή, γιατί υπάρχει αναβολή, Και το θέμα τη νομική βάση έχει απασχολήσει. Αυτό είναι το άρθρο 82, πράγμα που θέλαμε εμεί για την βάση τη δικαστική συνεργασία και επίση τεράστιε ανησυχίε για το τι μεταχείριση θα το θέμα. Ξέρετε ότι θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα αν ενταχθεί στην εσωτερική αγορά και η βάση είναι το 1.44 τη συνθήκη. αυτή είναι μια βασική μας ανησυχία, αλλά θέλω να ακούσω τι έχουν να πούν και οι συνάδελφοι. Εάν μπορείτε λοιπόν να μας πείτε περισσότερα από αυτού και πότε θα πρέπει να περιμένουμε την πρόταση πάω στους συντονιστές, η κυρία Μετσόλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, που ήρθατε σήμερα. Ε, σας ευχαριστώ για την ε, φανταστική σας Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα, τα οποία πρέπει να τα δούμε αμέσως, όπως είπατε και εσείς, στο χώρο των, της δικαιοσύνης και των ε, πολιτικών ελευθεριών. Αλλά σε αυτό το καθοριστικό σταυροδρόμιο για το για την πρόοδο του ευρωπαϊκού εγχειρήματο ε, νομίζω Πρέπει πάνω απ' όλα να βεβαιωθούμε ότι η δημοκρατία, το κράτο δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα γίνονται σεβαστά σε όλα τα κράτη-μέλη, στο καθένα ξεχωριστά από τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν τον περασμένο Οκτώβριο, Επίτροπε, εκφωνήσατε μια ομιλία στη Φιλανδία, νομίζω, ε, τονίσατε ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε κάτι για να ενισχύσουμε του μηχανισμού ελέγχου για το κράτο δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχατε απόλυτο δίκιο, διότι έκτοτε η κατάσταση έχει επιδεινωθεί στην ε, Μάλτα και τώρα στη Σλοβακία έχουμε δημοσιογράφους κατά τη διαφθοράς να δολοφονούνται. Αυτό δεν είναι τυχαίη φόνη, είναι βία η επίθεση κατά των μέσων μαζικής επικοινωνίας, της ελευθερίας της έκφρασης και ξέρουμε ότι δημοσιογράφοι δολοφονούνται ε, όταν το επιτρέπουν χαλαροί θεσμοί σε μια χώρα. Σε κάποια κράτη μέλη η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό που ενώ ε, οι μεταρρυθμίσεις ε, και όσα έγιναν στο κουτάκι του κατά λόγω ελέγχου είχαν το τικ που έπρεπε, ε, βλέπουμε στην πραγματικότητα να μην έχουν γίνει πραγματικέ αλλαγέ. Δηλαδή, επί χάρτη τα πράγματα έχουν μια μορφή και στην πραγματικότητα είναι τελείω ε, το αντίθετο αυτό που συμβαίνει. Αυτό ε, εντείνει τα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και δείχνει ότι πρέπει να αντιδράσουμε και να ανταποκριθούμε. Δεν συμβαίνει μόνο σε ένα κράτο μέλο μεμονωμένα. Είναι σαφέ ότι χρειάζεται όμω συγκεκριμένη ε, αντίδραση του μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να βασίζεται σε γνώση εμπειρογνωμόνων και να ελέγχονται όλα τα κράτη-μέλη εξονυχιστικά κάθε χρόνο. Όπως ε, ε, ο πίνακας αξιολόγηση, βαθμολόγησης μάλλον για τα θεμελιώδη δικαιώματα, είναι κάτι που πρέπει να ελέγχεται ανελαίητα και το ίδιο θα πρέπει να φροντίσουμε οι πολιτικοί να μην καλύπτουν απλώ τα συμφέροντα κάποιου. Θα κοιτάξετε να υπάρξει μια αναθεώρηση του μηχανισμού αυτού μέχρι το τέλο τη χρονιά όπω έχετε στο Ευρωκοινοβούλιο. Συνάδελφοι, να θυμίσω ότι υπάρχει και μια αντιπροσωπεία Κοντ Λιμπ μεθαύριο. Θα υπάρξει επίσκεψη. Νομίζω ότι είναι μια ε, αρκετά έγκαιρη και εύστοχη αντίδραση τη Επιτροπή μα, η κυρία Σίπελ από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Επίτροπο Γιούροβα που έθιξε τόσα πολλά σημαντικά ζητήματα που είναι μέρο του χαρτοφυλακίου τη. Και μα καλούν να θέσουμε κι εμεί μια σειρά από ερωτήσει. Θα ήθελα να κάνω 4-5 παρατηρήσει και να ξεκινήσω και πάλι με το κράτο δικαίου. Πιστεύω ότι επί χρόνια αυτό είναι μια απέτηση του Κοινοβουλίου που επαναλαμβάνεται και ουδέποτε λάβαμε σαφή απάντηση για το πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση. Η Ρομπέρτα Μετσόλα ήδη ανέφερε τη Μάλτα και τη Σλοβακία, αλλά για να είμαι και ειλικρινής, νομίζω μακροπρόθεσμα οι εξελίξεις στην Πολωνία είναι επίσης ανησυχητικές. Ε, δεν βλέπω γιατί το Συμβούλιο ε, δεν ε, κάνει κάτι για το άρθρο της κατεπήγουσας ε, διαδικασίας. Θα πρέπει να γίνει μια συστηματική διαδικασία μεταξύ φίλων, να προειδοποιεί ένα στον άλλο ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Η κατάσταση επιδεινώνεται μάλιστα, εάν σκεφτούμε και τι γίνεται στην Ουγγαρία, διότι ουδέποτε μπορέσαμε επισήμω να εκφράσουμε τις σοβαρές μας ανησυχίες, ε, κάτι που πραγματικά ισχύει όταν αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τι θα γίνει λοιπόν, τι προετοιμάζετε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Πιστεύετε ότι χρειαζόμαστε ως Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερες εξουσίες για να έχουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, μια γρήγορη και ταχεία αντίδραση ε, από την πλευρά των κρατών μελών όταν υπάρχουν τέτοια θέματα. Έπειτα να περάσω, και αυτό δεν θα σας εκπλήξει, στην ε, ασπίδα της, ε, του ιδιωτικού βίου. Πολλοί είναι οι φορείς που έχουν εκφράσει επικριτικές παρατηρήσεις και ενδιασμούς λόγου χάρη για τον ε, ε, διαμεσολαβητή άντρα ή γυναίκα γιατί η ομάδα εργασία του άρθρου 29 είπε ότι αυτό ακόμη δεν μπορεί να προβλεφθεί και θα πρέπει να προβλέψουμε τα κατάλληλα ένδικα μέσα πριν από ένα δικαστήριο. Αλλά πρέπει να οριστεί και μια προθεσμία που είναι 28, 28 Μαΐου πριν ε, προσφύγουν στα εθνικά δικαστήρια και το θέμα να απευθύνει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο οι φορεί τι βήματα σε σχέση με αυτή τη διαδικασία προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Έχετε την πεποίθηση ότι η προθεσμία της 25ης Μαΐου θα γίνει σεβαστή. Ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τον ιδιωτικό βίο είναι το τμήμα 7 που επετράπη ξανά ε, στις Αμερικανικές αρχές ώστε να παρακολουθούν ουσιαστικά ε, δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών. Ποια είναι η εξαλογισή σας για αυτήν την ε, προεξουσιοδότηση για την ασπίδα ιδιωτικότητα για το ΦΙΖΑ. Και δύο-τρει σύντομε ερωτήσει για το Μετρό Επιβατών. Ποιε είναι οι συνέπειες; της ε, ε, απόφασης του για το ε, Ευρωπαϊκό PNR, Μητρό Επιβατών και τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση του πολυεναμενόμενου Ευρωπαϊκού PNR και για τον GDPR. Να πω ότι βλέπω να υπάρχουν πολλά κενά, πολλά παραθυράκια για τα κάτι μέλη να το εφαρμόσουν όπως θέλουν. Οπότε η ερώτησή μου είναι, Είστε έτοιμοι να περάσετε σε διαδικασίε που παραβάσει αμέσω κατά των κατομελών, εφόσον δεν έχουν απαντήσει εγκαίρως ε, στην εφαρμογή των μέτρων. Για το GDPR. Είναι και το θέμα των ε, προσώπων μικρών επιχειρήσεων που δεν είναι έτοιμοι ακόμα. Οπότε, αν θέλετε να μας πείτε κάτι και γι' αυτό, διότι πιέζει ο χρόνος και τα εθνικά κοινοβούλια μας περιμένουν σε συνάντηση είναι ένα σημείο που απασχολεί τα κράτη-μέλη. Για του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ, η κυρία Στίβεν δεν είναι εδώ, αλλά κυρία Γιούρεκ, θέλετε εκ μέρου των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών να μα πείτε κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο κύριο Γιούρεκ, ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε που ήρθατε στην Επιτροπή μας. πάντοτε να συζητάμε το εκτό τη πολιτική τη Επιτροπή είναι θετικό. Έχω τι εξή ερωτήσει. Πρώτον, η τοποθέτηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την άμεση δημοκρατία. Η Ρουμανία τώρα προετοιμάζει ένα δημοψήφισμα Σαν αυτόν τον ορισμό της ε, οικογένειας, κάτι το οποίο πρόκειται να ενταχθεί μετά στο Σύνταγμα της χώρας. Σχεδόν ένα εκατομμύριο Ρουμάνων ζήτησαν να γίνει η σχετική αλλαγή. Πάντως τώρα πολλοί πολιτικοί θέλουν να θαυτεί το θέμα για να μην ε, γίνει το δημοψήφισμα. Καταλαβαίνω ότι εσείς δεν ε, θα παρέμβετε, αλλά είμαι περίεργος για το πώς βλέπετε τα πράγματα. Ο κόσμος θέλει την αλλαγή σε αυτό το θέμα. Και τι θα συμβεί. δεύτερη ερώτησή μου. Για τα θεμελιώδη δικαιώματα και το πώς προσεγγίζει η Επιτροπή τον ρόλο των γονέων σε ανατροφή των παιδιών. Γνωρίζουμε ότι ο χάρτη των δικαιωμάτων στο άρθρο 14 ορίζει τα των σχετικών δικαιωμάτων των γονέων και θεωρεί ότι αυτό είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα των γονέων. Δηλαδή να ανατρέφουν τα παιδιά τους όπως θεωρούν σωστό. Κύριε Επίτροπε, ήδη μας αναφέρατε κάποιες προσδοκίες που έχετε όσον αφορά τους ΛΟΑΔ. Άρα, πώς προσεγγίζεται το θέμα σε σχέση με τον ορισμό που θα πρέπει να εισαχθεί στην ε, διδακτή αίλη των σχολείων για το τι θα πει η οικογένεια. Δεν έχουμε εδώ και θέμα δικαιωμάτων της μειοψηφίας. Για την ε, Άλντε η Σοφή Νετφέλτ. Χαίρομαι που όλα και περισσότερες ε, χώρες προβληματίζονται ότι δεν είναι υπόθεση της κυβέρνησης το ποιον μπορεί να αγαπήσει, να παντρευτεί κανείς, να κάνει παιδιά. Και άκουσα επίσης η Ρομπέρτο Μέτσολα για το 702, το PNR, το Συμφωνία DRF και είχαμε απευθύνει μια επιστολή για την πρόταση των ΙΠΑ, ούτως ώστε να υπάρχει ένα εθνικό κέντρο διαλογής και ελέγχου και οπότε θα υπάρχει μια διασύνδεση των βασικών δεδομένων των δεδομένων που θα περιλαμβάνει και δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών. Ε, αυτό αντιβαίνει σε πάσα συμφωνία που έχουμε ε, συνάψει με τις ε, ΗΠΑ που έτσι να το πω διπλωματικά δεν είναι και τόσο νομικά στεγανές οπότε ε, εσείς προτίθεστε να είστε αποφασιστικοί ως προς τις ΗΠΑ είπατε κάτι τέτοιο, αυτό θα ήταν πάρα πολύ θετικό. Ε, πάντως τα τελευταία 15 χρόνια μάλλον ε, χαλαρή ήσασταν στην αντιμετώπιση των Αμερικανών για αυτά τα θέματα. Τώρα κάτι άλλο το οποίο το έχουμε ξαναπεί με σας. Τι γίνεται με τον προϋπολογισμό, τι γίνεται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, γιατί ξέρετε προβληθίζομαι ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής ε, δεν θέλουν να υπάρχει αυτή η ένδειξη στον προπολογισμό του litigation fund αυτού του Ταμείου Επίλυσης Ενδικών Διαφορών. Είναι θέμα αξιοπιστίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μιλούμε για τον ρόλο σας ως ε, φύλακα των συνθήκων και κυρίως για το θέμα της δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μα είναι πολλοί οι Ευρωπαίοι οι οποίοι νιώθουν ε, απογοήτευση σε σχέση με τον διορισμό του νέου ναι, Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εγκρίθηκε από το Σώμα των Επιτροπών. Και ο κύριο Ζελμάιερ έχει τα δικά του σχέδια και προσωπικά και για την νομική υπηρεσία τη Κομισιόν. Και μου στέλνει κόσμο email και μου λέει, Μα πώ εγώ να εμπιστεύομαι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όταν ενεργεί κατά τον τρόπο το πιο ισχυρό θεσμικό όργανο. Θα ήθελα να καταλάβω Μα πώς εδώ να είμαστε αξιόπιστοι, ε, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι μόνο ω διοίκηση, αλλά ως πολιτικό όργανο, δηλαδή το Σύνολο των Επιτρόπων. Πω, από ποίου που ενέκριναν αυτόν τον διορισμό, πώς έγινε κάτι τέτοιο. Ο Πρόεδρο. Και η Κονιλία Ένστη για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Παρακολουθώ αυτό που μας είπατε, αυτό που έχουμε να συζητήσουμε. Έκαναν κάποια σχόλια βέβαια και οι συνάδελφοι. Διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διαλύεται, δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις, ενώ έρχομαι τις ΗΠΑ από την άλλη πλευρά που μας παρουσιάζουν μια τελείως διαφορετική κατάσταση με έναν ε, εμπορικό πόλεμο και την εισαγωγή των δασμών που επιβάλλονται από πλευρά των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Ε, άρα λοιπόν το ερώτημα είναι τι πρόκειται να διαπραγματευτείτε, τι μπορείτε να διαπραγματευτείτε για, τον, ε, ε, για το σύστημα προστασίας προσωπικών δεδομένων, πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση, τι μπορούμε να περιμένουμε. Ε, τρέφω άπειρο, άπειρα αισιοδοξία και βλέπω ότι είναι καθόλου ικανοποιητική αυτή η κατάσταση. Το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Πολύ ωραία. Στις 25 Μαΐου λέτε θα τεθεί σε εφαρμογή σε όλα τα τμήματα ο κανονισμός και το e-privacy, ηλεκτρονικό η προστασία του ιδιωτικού βίου και ε, η ισχύση του κανονισμού για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη και τα θεσμικά όργανα. Αυτό που εμείς ζούμε όμως, και μπορώ να το πω τουλάχιστον προσωπικώς από το τελευταίο διάστημα, το Συμβούλιο έχει παρεμποδίσει κάθε εξέλιξη ε, και από ό,τι φαίνεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων θέλει να την ε, εγκαταλείψει τουλάχιστον για ορισμένου τομεί ή να την παραβλέψει. Ειδικά για τη Europol, παραδείγματι. εσεί ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις προτάσεις μας πώ θα σχεδίσετε τα θέματα των ε, ε, αποκεντρωμένων υπηρεσιών και δι' αυτών που έχουν να κάνουν με την επιβολή του νόμου και ε, ε, εάν θα ακολουθήσετε τη λογική που λέει ότι πρέπει και αυτέ να τηρούν την κανονισμό για των προσωπικών δεδομένων, ή αν θα ακολουθήσετε τι επιλογέ του Συμβουλίου που παρεμποδίζει αυτή την ε, εξέλιξη, θα υπάρχει η δυνατότητα να ταθεί σε εφαρμογή εγκαίρω και πλήρω ο κανονισμό, ή θα είναι ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση. Γιατί θεωρώ ότι εδώ έχει κατακαιρματιστεί κάθε, έχει καταποντιστεί κάθε έννοια εμπιστοσύνης μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο βλέπουμε ότι ακολουθεί παρελκυστική πολιτική, προσπαθεί να αποκλείσει από κάποιους τομείς ιδιαίτερα την εφαρμογή και επιβολή του νόμου, ε, τον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για το άλλο θέμα που αναφερθήκατε, διακρίσεις στα παιδιά Ρωμά, ένα θέμα που έχουμε συχνά συναντήσει, κριτήσεις, στρατηγικές για την ενσωμάτωση, που θα επαληθευθούν τον ε, το φθινόπωρο, πολύ καλά, αλλά δεν αρκούν όλα αυτά. Έχετε υπόψη κάποια πιο σκληρά μέτρα που θα μπορούσατε να απαιτήσετε, γιατί είναι σκανδαλώδης ο τρόπο με τον οποίο ε, υφίστανται διακρίσεις εις βάρος τους η Ρωμά. Και αντί για πρόοδο διαπιστώνουμε σε ορισμένα κράτη ακόμη και οπισθοδρόμηση. Έτσι λοιπόν μπορεί να αναλυφθούν πιο σκληρά μέτρα ή θα τα αφήσετε στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών. Η κυρία Σαρζεντίνη για τους πράσινους. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ξεκινώ ευχαριστώντας την Επίτροπο για τα νέα μέτρα υποστήριξης ε, των ΛΟΑΔΜΑ και βέβαια όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών, στην καταπολέμηση της ρητορικής μίσου, στη δυνατότητα και μόνο να γίνεται διάλογος για τα θέματα γάμου ε, ομοφιλοφίλων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η δυνατότητα και χαιρόμαστε ιδιαίτερως που πιέζεται για να προχωρήσουν αυτές οι προτάσεις. Ένα άλλο θέμα για την καταπολέμηση των διακρίσεων, στο οποίο ωστόσο έχουμε δυσκολίες, ε, τόσο εμείς όσο και η Επιτροπή, ε, θέλω να αναφέρω την ε, εγκάρσια οδηγία για την ισότιμη μεταχείριση. Δεν έχω ακούσει κανείς να το συζητάει από το 2009 μέχρι τώρα το θέμα αυτό. Βλέπετε κάποια κινητικότητα σε επίπεδο συμβουλίου και υπάρχει κάτι που μπορούμε εμείς μαζί σας να ε, αναλάβουμε ω πρωτοβουλία. Ένα άλλο θέμα, τα δικαιώματα των θυμάτων, η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων. Έγινε διαπραγμάτευση το 2011 ολοκληρώθηκε το 2012 η επεξεργασία Το 2015 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε όλα τα κράτη-μέλη μεταφορά τη οδηγία σε εθνικό δίκαιο. Ωστόσο αυτό δεν έχει συμβεί και φαντάζομαι ότι και εσεί ανησυχείτε όπω και εμεί. Έχετε υπόψη κάποιε διαδικασίε προσφυγή ε, για παράβαση τη συνθήκη ή έχετε ενδεχομένω ξεκινήσει κάποιε και κάτι ακόμη που απασχολεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχετε κάποια γενική εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη μεριμνούν ώστε να μην υπάρξει διάκριση μεταξύ των θυμάτων που έχουν ε, τα σχετικά αποδεικτικά επί, τα σχετικά ε, στοιχεία ταυτότητα, τα χαρτιά δηλαδή όπως γνωρίζει το άρθρο 1 και εκείνων που δεν ε, έχουν νομιμοποίηση διαμονής. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα πρέπει οπωσδήποτε να το προγάγουμε και θέλω περισσότερες πληροφορίες από σας αν έχετε. Επίσης ευχαριστώ πολύ για τα συγχαρητήρια που δώσατε στο Κοινοβούλιο για την οδηγία για την καταπολέμηση νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Αυτό το οποίο έχουμε επιτύχει και σε συνεργασία με την Εστονική Προεδρία βεβαίω πιστεύω είναι σημαντική πρόοδος. Ωστόσο υπάρχουν τα οποία δεν έχουν και ξέρω ότι έχετε αποστείλει επίστολες σε μια σειρά από αυτά τα κράτη-μέλη, προχωρήσει στην υλοποίηση της οδηγίας και ε, διερωτώ αν έχουμε περάσει σε μια επόμενη φάση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα εργαλείο για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να θέλουν να το, να το προωθήσουν και με απογοήτευση βλέπω ότι υπάρχουν κράτη συμπεριλαμβανωμένοι οι σκητιστικοί μου πατρίδες των κάτω χωρών που δεν έχουν ακόμα προχωρήσει, υλοποίηση ούτε τις ε, προηγούμενες οδηγίες, πόσο δε μάλλον τις ε, επόμενες. Στο νομικό πλαίσιο επίση που ξεκινάει αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή κυρία Επίτροπε, μπορούμε να περιμένουμε κάποιες συστάσεις, κάποιες προτάσεις για αιρεσιμότητα σε σχέση με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, η οποία θα στηρίζεται στις αρχές του κράτους δικαίου, γιατί πολύ είναι η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία φτάνει σε κράτη-μέλη με ε, σχετικά ευέλικτη ανάγνωση των όρων του κράτους δικαίου. Μήπως ήρθε η ώρα να ανοίξει και αυτή η συζήτηση. Μπορούμε να περιμένουμε τέτοιες προτάσεις στο εγγύς μέλλον. ευχαριστώ. Η κυρία Κοράτσα Πρόεδρε, ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την πρωτοβουλία και την προσήλωση στην καταπολέμηση του ε, διαδικτυακού, του διαγραμμικού παράνομου περιεχομένου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως άλλωστε και το θέμα της προστασίας από σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και διαγραμμικά. Έχετε λοιπόν κάνει μια ριζική ε, προσέγγιση και σε συνεργασία με, την, ε, ε, με τις επιχειρήσεις που μπορεί να έχουν επιτρέψει τη διακίνηση τέτοιου παράνομου υλικού που αφορά παιδιά. Επίσης, σε σχέση με τη σύμβαση την προηγούμενη εβδομάδα, ο Πρόεδρος Ταγιάννη κήρυξε το ε, την έναρξη της Ολομέλειας με απερίφραστη τοποθέτηση για τη σύμβαση. Διαρωτώ λοιπόν πώς έχουν προχωρήσει τα θέματα αυτά. Έχει ολοκληρώσει το Συμβούλιο τις εργασίες για την πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύμβαση, στη σύμβαση και επίσης έχουμε ζητήσει να αναλυφθεί διάλογος από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν επιφυλάξει, δεν έχουν κυρώσει κτλ. Και Γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια μέλη τα οποία έχουν παγώσει διαδικασίε κυρίω. Ακόμη και η Προεδρία αυτή τη στιγμή, η Βουλγαρική, στα θέματα που αφορούν ιδιαίτερα την ε, βία με βάση το φύλλο και την μεταχείριση των φύλων. Παρακαλώ λοιπόν να ασκήσετε κάθε πίεση στην Προεδρία στην Βουλγαρία συγκεκριμένα στο θέμα αυτό να μπει στην διάρκεια του εξαμήνου τη στην ε, ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου. Επίσης ο κανονισμό για την προστασία του προσωπικού βίου ιδιωτικού βίου. Συνεχίζεται η συζήτηση του θέματος αυτού. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε τις βέλτιστες δυνατέ τις καλύτερες δυνατές ε, προδιαγραφές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, χωρίς όμως να υπονομεύσουμε την καινοτομία και με ασφάλεια δικαίου, μια νομοθεσία δηλαδή η οποία θα είναι σύμφωνη με το γενικό κανονισμό, αλλά ταυτόχρονα και δεν θα παρεμποδίσει την ε, τεχνολογική εξέλιξη. Και επίσης συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που μας ανακοινώσατε ώστε ε, να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ. Λυπούμε και εγώ διαπιστώνω που, ότι η οδηγία για την αντιμετώπιση των διακρίσεων εις βάρος των ΛΟΑΔΜ έχει παγώσει σε επίπεδο Συμβουλίου και σας παρακαλώ να μας πείτε τι μπορείτε να κάνετε προκειμένου να την ε, απεμπλέξετε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρεβόνταλόν Πονφά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Πίτροπε, όπως είπε και η συνεισηγήτρια και συνάδελφος ε, για την υπογραφή της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω και εγώ να το θίξω αυτό το θέμα, διότι θα χρειαστούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα, για το εξή. Μπορείτε να μα πείτε τι υπόθηκε στην συνεδρίαση τη ομάδα εργασία ε, ε, στο Συμβούλιο στι 26 Φεβρουαρίου για τον κώδικα συμπεριφορά, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και ένα θέμα για το οποίο έχετε την πλήρη υποστήριξή μα σε ό,τι αφορά αυτή τη νομική μάχη η οποία ε, μένεται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Συμβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για να δούμε αν είναι αρμοδιότητα ή όχι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω ε, ξέρετε και εμεί ζητήσαμε από την νομική υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου την δική του έμπειρη γνωμοσύνη και επιβεβαίωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διατηρήσει μια αρμοδιότητα γενικότερη από αυτήν που αυτή τη στιγμή αμφισβητούν κάποια από τα κάτι μέλη στο Συμβούλιο. Πώ βλέπετε να δημορφώνονται τα πράγματα, το είπε και η συνάδελφο Άννα Μαρία Κορατσαμπίλτ με τη Βουλγαρία που αυτή τη στιγμή έχει εγκαταλείψει τη δέσμευση για την υπογραφή και την κύρωση από πλευρά τη ίδια τη Βουλγαρία τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη έχει την Προεδρία του Συμβουλίου. Θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο ερχόμενο εξάμεινο για το σκέλο αυτό που είναι ε, άκρα σημασία. Ευχαριστώ για αυτή την πολύ χειροπιαστική και συγκεκριμένη απάντηση. Ευχαριστούμε κυρία Κιέγγε. Ευχαριστώ Επίτροπε. Την περασμένη εβδομάδα το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε την έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2016. Η έκθεση αυτή καταγράφει και το γεγονός ότι εντός των 100 μελών το φαινόμενο της διακριτικής μεταχείρισης δυστυχώς εντείνεται. Είναι σε φάση εντατικοποίησης από πολλά κράτη-μέλη. Ιδίως ό,τι αφορά κάποιες κατηγορίες πολιτών, ε, σε ό,τι αφορά τους μετανάστες, ε, σε ό,τι αφορά τους Ρωμά, ήδη εφήγει αυτό, σε ό,τι αφορά τους μετανάστες πιο συγκεκριμένα για τους ε, αφρικανικής προέλευσης μετανάστες. Αυτό βλέπουμε βλέπουμε να ανησυχεί πολύ και με τον πυροβολισμό στην Ματσεράτα ορισμένων ε, πολιτών πριν από λίγες εβδομάδες όπου δέχτηκαν πυροβολισμούς ε, κάποιοι Αφρικανοί όλοι αφρικανικής προέλευσης ε, με την προσπάθεια να υπάρξουν όλο, όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα. Εδώ λοιπόν ε, ελεύθεροι σκοπευτέ χτυπήσανε πλήθος προκειμένου να χτυπήσουν ε, Αφρικανούς. Ποια θα πρέπει να είναι η νομική μα απάντηση, τι μπορούμε να κάνουμε για να υπάρξει μια στρατηγική σε όλα τα κράτη-μέλη. Θελήσαμε να υπάρξει ένα Ευρωπαίο συντονιστή για την καταπολέμηση τη ξενοφοβία. Αυτό αναφέρεται και στην έκθεση που υιοθετήθηκε. Και μια ευρωπαϊκή στρατηγική σε ό,τι αφορά ορισμένε Ορισμένε αντιδράσει στην Ισλαμοφοβία, ε, στους, ε, στα προβλήματα από τους Ρωμά, ε, στις εκφράσεις μίσου, Επίτροπε, σκοπεύετε να ακολουθήσετε αυτήν την κατεύθυνση σε ό,τι αφορά και την αφρικανοφοβία και ήθελα να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θα δεχτεί το αίτημά μας για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για την καταπολέμηση των ε, φοβικών ε, συμπεριφορών και την πρόθεση των δικαιωμάτων των πολιτών. Θα σταθούμε ε, στο πλευρό της κοινωνίας των πολιτών σε όλα αυτά. Ευχαριστούμε Ιάννα Χέτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο γιατί πάντοτε είναι πρόθυμη να έρθει και να απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Θα ήθελα να της απευθύνω ένα συγκεκριμένο ερώτημα για την οδηγία, την οριζόντια οδηγία για την ισότητα των ευκαιριών. και πέραν αυτής και για την οδηγία κατά της εμπορίας ανθρώπων που θα έπρεπε να διαθέτει επίσης ε, να προσεγγίζεται και με μια διάσταση ισότητας των ε, φίλων ίσων ευκαιριών. Στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων βλέπουμε ότι διαρκώς χρειάζεται να εξεύρουμε νέες λύσεις γιατί αλλάζουν οι μορφές στο φαινόμενο αυτό. Η Επίτροπος είπε ότι θα υποβληθεί ε, θα δημοσιευτεί ανακοίνωση για την καταπολέμηση της εμπορίας των ανθρώπων. Εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο θέλουμε να καταρτήσουμε την στρατηγική μας καθώς το φαινόμενο αυτό μεταβάλλεται διαρκώς ο τρόπος που οι έμποροι ανθρώπων ε, ε, οργανώνονται, αλλάζει συνεχώς Το ερώτημα λοιπόν είναι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβλέπει τις ανάλογες προσαρμογές στην πρόταση οδηγία. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μετσόλα θέλει πάλι το λόγο. Ναι, με συγχωρείτε πρόεδρε. Μετά το θέμα αυτό για τους Αφρικανούς ε, και η συνάδελφο μου ζήτησε να θέσω το ερώτημα για τη στρατηγική κατά τον Ρωμά, ε, μάλλον υπέρ των Ρωμά μετά το 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώ αποτιμά τώρα την ένταξη των Ρωμά, τι βήματα προβλέπει να κάνει από το 2020 και μετά και πώς σκοπεύει να αναβαθμίσει το πλαίσιο για το διάστημα μετά το 2020 όπω ζητάτε από το ψήφισμα που πρόσφατα ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο. Και τα τι δαπάνε έγιναν από το 2011, ποια είναι η κατάσταση μετά Δυτικά Βαλκάνια και την διαδικασία προσχώρησή του, καθώ και του Ρωμά, και πώ θα υπάρξει καλύτερη παρακολούθηση. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Διαθρωμένο διάλογο ονομάζεται, αλλά δεν ήταν τόσο διαθρωμένο. Μπίργκιτ, έχει κι ερώτηση. Χάνουμε τελείω τη διάρθρωση. Ναι, εντάσσεται στην όλη διάρθρωση. Ξέχασα να θέσω ερώτηση για το GDPR τα συζητήσαμε δια μακρόν, δια μακρότατον και θα έπρεπε να δούμε ότι παρά τι ανησυχίε που είχαν εκπαιδευτεί εδώ στην Επιτροπή μα, λίγε εβδομάδε πριν αρχίσει να εφαρμόζεται, το Συμβούλιο αρχίζει να περνάει σε κάτι διορθωτικά. Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ ω τώρα κάτι τέτοιο. Ε, τι διορθωτικά είναι αυτά, τι γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι θα ε, ε, επιφυλάξει αυτό για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι στρατηγική ακολουθεί αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο. Ναι, διορθωτικά του Συμβουλίου λέτε. Η απάντησή μου εμένα θα ήταν οπωσδήποτε ναι. Ναι, οπωσδήποτε. Τόσα πολλά ερωτήματα σας τέθηκαν. Κανένα εκατομμύριο ερωτήσεις. Μαζέψου. Τα περισσότερα όμω άπτονται του χαρτοφυλακίου σας, οπότε παρακαλώ όσο καλύτερα μπορείτε απαντήστε. Ευχαριστώ, λέει η κυρία την επόμενη φορά θα πρέπει να έχουμε ε, κάπως πιο, πιο στενό πεδίο συζήτησης, αλλά να προσπαθήσω, να προσπαθήσω να καλύψω τις ερωτήσεις. Πρώτα πρώτα, μας είπατε για την ε, νομική βάση και να σας πω το χρονοδιάγραμμα την πρόταση θα την εγκρίνουμε τον Απρίλιο. 17 Απριλίου λέμε τώρα. Μα ήδη έχει αναβληθεί πολλές φορές. Γιατί, γιατί ήταν περίπλοκο, ήταν ε, ένα σωρό θέματα εδώ πάρα πολύ επίμαχα, λεπτά. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και επιλύσουμε. Οπότε έχουν το άρθρο 82 για την δικαστική συνδρομή στα ποινικέ υποθέσει κλπ. Επίση, είπαμε ότι θα πρέπει να κάτσουμε και να εξισορροπήσουμε. Να υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό εργαλείο. Να βοηθούν δηλαδή οι διεκτικέ αρχέ να έχουν τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζονται διασυνοριακά. Κάτι που τώρα δεν το έχουν. Και Όλα αυτά μέσα σε ένα πεδίο ξεκάθαρο. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα και όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία. Τέτοιο παιδί εφαρμογή θέλουμε και τέτοια βάση. Επομένως να είναι εύχριστο φιλικό στη χρήση αυτό το εργαλείο. και επίσης να μπορούμε να συντονιστούμε με τις ε, εταιρείε πληροφορικής στις οποίες θα απευθυνθούν οι διοκτικές αρχές και να είναι σύνομα τα σχετικά αιτήματα. Οπότε έτσι θα πρέπει να επιζητηθεί μια δόκιμη λύση για κάτι το οποίο θα αφορά και τις τρίτες χώρες. Τα είπαμε όσον αφορά τους ε, Αμερικανούς εταίρους μας για το καθεστώς αμοιβαιότητας. Πώς δηλαδή θα βρούμε την καλύτερη των λύσεων, μια που διαπιστώνουμε ότι πρώτα φορά πρέπει να διαβιβάσουμε από τι δικαστικέ ΗΠΑ, όπου θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι διοικητικέ αρχέ μπορούν να έχουν αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία. Και όλα αυτά με κάποια ισόρροπη μεταχείριση, δίκαιη μεταχείριση. Δηλαδή, εφαρμογή του νόμου και προστασία όμως του ιδιωτικού βίου και των δικαιωμάτων. Τώρα πάλι για την πληροφορική, γιατί προφανώς δικαστές και εισαγγελείς θέλουν να έχουν τέτοιο εργαλείο στα χέρια τους. Και οι ίδιες ε, οι τρεις πληροφορικής θέλουν ασφάλεια δικαίου, θέλουν πιο στεγανούς κανόνες, θέλουν να είναι ξεκάθαρο το τοπίο για το τι θα πρέπει να κάνουν σε κάθε περίπτωση όταν απευθύνονται σε αυτές οι ιδιωτικέ αρχές για e-evidence, για αυτά τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Οπότε εμείς πασχίζουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις προτάσεις ε, Λαμβάνομαι υπόψη ε, το ότι εσείς παρακολουθείτε το τι γίνεται, ελέγχετε για τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε και για το μέλλον όσον αφορά αυτόν τον έλεγχο. Μα όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Χρειαζόμαστε αυτή την νομοθεσία. Είναι θέματα ποινικής δικαιοσύνης, αλλά ακόμα εκκρεμούν πολλά ερωτηματικά και ελπίζω θα τα πάμε καλά. Έχουμε αρχίσει τη συνεργασία με του Υπουργού Δικαιοσύνη από το 16, αν δεν κάνω λάθο, που είχαμε την Ολλανδική Προεδρία και εκείνοι και οι Υπουργοί Δικαιοσύνη ανυπομονούν. Άρα, μετά από όλε αυτέ τι συζητήσει, κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Για το PNR τώρα, και αυτό που ζήτησε η κυρία, ρώτησε κυρία Σίπελ, όσον αφορά την απόφαση του ΔΕΚ, όσον αφορά τις τρίτες χώρες. Ε, βέβαια, είναι φανερό ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανακαθορίσει την προσέγγιση της όσον αφορά τις συμφωνίες PNR πριν, πριν μάλλον συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Μια που προκειμένου έχουμε το θέμα των σχέσεων με το Μεξικό. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει πριν να αρχίσουμε συνομιλίες με άλλες τρίτες χώρες. Όπως γνωρίζετε <clears throat> η, ε, η Ιαπωνία καίγεται για να τα συζητήσουμε εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων. Άρα είναι καυτό το θέμα. Και θα συνεχίσουμε να εξηγούμε στους διεθνείς εταίρους για το τι νομικό πλαίσιο υπάρχει για τη διαβίβαση δεδομένων PNR και θα αναδεικνύουμε πάντοτε ότι πρέπει να βελτιώνουμε τα της ασφαλείας υπέρ των συμπολιτών μας και, αλλά ταυτόχρονα και να προστατεύουμε τα προσωπικά τους δεδομένα. Και νομίζω ότι σαφώς έχει προκύψει πώς θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες από διάφορες συμφωνίες Πάντως το δικαστήριο έκρινε τα της ανταλλαγής δεδομένων με τον Καναδά. Το θέμα έχει πάρα πολλές νομικές πλευρές, τεχνικές νομικές πλευρές, τέλος πάντων το επεξεργαζόμαστε με τους ε, συναδέλφους για το PNR. Αυτά όσον αφορά τώρα το θέμα της προστασίας του ιδιωτικού βίου, privacy, ναι, ναι, ναι. Όπως είπα θα είμαι σκληρή αυτή τη φορά. Και όπως είπαμε και την τελευταία φορά πήγα και τα είπαμε τον Μαρτίο για τις δυσκολίες που υπήρχαν με την καινούργια κυβέρνηση αλλά έχω πει από πολλά βήματα ότι η δική μας θέση έχει θεμέλιο την εμπιστοσύνη, τις ε, δεσμεύσεις μας Άρα είναι θέμα δικό μας αλλά και δικό τους των Αμερικανών. Ήταν ξεκάθαρο σε αυτές τις ε, συστάσεις της ομάδας εργασίας 29. Εγώ για την προθεσμία θα το επισημάνω σε όλους στους οποίους πρέπει να το επισημάνω. Ήδη Πάντως κάποιες συστάσεις μας τις έχουν δεχθεί. Για την πιστοποίηση, για την επισήμανση όσον αφορά τα force claims, Πάντως εμείς θέλουμε να λειτουργεί με πλήρες αρμοδιότητες η υπηρεσία του διαμεσολαβητή της διαμεσολαβήτριας. Αυτά έχουν προτείνει και οι Αμερικανοί. Θεωρούν ότι ε, ε, εκεί θα πρέπει να υπάρχει η αρμοδιότητα ε, γιατί πρόκειται για ανεξάρτητη υπηρεσία στην Αμερικανική κυβέρνηση και εκείνοι θα διεκπεραιώνουν τις καταγγελίες μας όταν θεωρούμε ότι οι διοικητικές αρχές υπερβαίνουν τα της αρμοδιότητός τους για τα δεδομένα και ότι ενεργούν τέλος πάντων εκτός της νομιμότητας. Επίσης Είπαμε ότι θα πρέπει κάποιο να έχει πλήρη απασχόληση ως διαμεσολαβητής ή διαμεσολαβήτρια και είπαμε ότι σε αυτό είμαστε υποχώρητοι. και για την Σχετική Επιτροπή αλλά και για άλλους διορισμούς συναφών αρμοδιτών. Και όταν πήγα εκεί ε, είπαμε ότι το Privacy Shield δεν είναι υψηλή προτεραιότητα αυτή η ασπίδα ιδιωτικού βίου. Ναι και είπαμε ότι θα καταστεί προτεραιότητα ξεκαθαρίζοντας ότι εμείς εάν δεν υπάρχει το privacy shield θα τραβήξουμε το χειρόφρενο. Θα σταματήσουμε τη συνεργασία. Θα κλείσουμε τις για στο σύστημα. Γι' αυτό θέλουμε να καλύπτει τις επιχειρήσεις και των δύο πλευρών χρειάζεται να υπάρχει μια σχετική νομική ρύθμιση. Εξαντλείται η υπομονή μου. Και είμαστε ξεκάθαροι σε σχέση με αυτό το σημείο. Όταν δε πάω στην Washington θα έχω την ε, νομική ανάλυση για το τι ισχύει σχέση με το 702 και για τις συνέπειες της νέας Αμερικανικής νομοθεσίας. Θα ζητήσω ενδελεχή νομική ανάλυση Τι εγγυήσεις που υπάρχουν από πλευρά της Αμερικής. Όσον αφορά τις ε, πολιτικές οργανώσεις, τι γίνεται σχετικά με τις εποπτικές αρχές, και τι, τι λένε και οι επιχειρηματίες επίσης. Ναι, θα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί, σκληροί και να τηρηθούν οι προθεσμίες επακριβώς. Αυτό αφορά και την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου. Είναι πολύ ε, σημαντικά και τα σχετικά με αυτήν την Επιτροπή. Τώρα για το κράτος δικαίου για να δούμε τι ρωτήσει Ναι, θα πρέπει το πλαίσιο αυτό να θωρακιστεί και θα πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσουμε περισσότερο τι εννοούμε για την αρχή του κράτους του δικαίου. Μα είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας. Και εκεί θα πρέπει να βασίζεται κάθε δημοκρατικό κράτος. Προς έκπληξή μου. Πολύ. Και επίσημη πιστεύουν ότι αν κάποιος κερδίσει τις εκλογές, τότε κάνει ό,τι θέλει. Μα δεν προβλέπει κάτι το κράτος δικαίου. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η διέρωση των εξουσιών είναι κάτι που η πολιτική εξουσία δεν θα πρέπει να θίξει. Βεβαίως, η κάθε χώρα έχει τα δικά της θα πρέπει όμω να επαγγελματούν περισσότερο για το κράτο δικαίου και πάντοτε ακούω τα ίδια και τα ίδια. Το ίδιο επιχείρημα ότι υπάρχουν διαφορετικά συστήματα, υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν υπάρχει στεγματικό δικαστήριο, ε, κάποια κράτη που δεν υπάρχει δικαστικό συμβούλιο, ανώτο δικαστικό συμβούλιο. Ε, ωραία, εντάξει, εμεί έχουμε ένα σώρο συστήματα. Αλλά θα πρέπει όλα και το καθένα να αποδίδει, να, να, να, να τηρεί, να συμβαδίζει με το κράτος δικαίου. Και εμείς θα πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε ακριβώς τι εννοούμε στην Ένωση με το κράτος δικαίου. Δηλαδή, ε, τι θα κάνουμε τα δεδομένα, τι μηχανισμούς θέλουμε, πώς θα έχουμε καλύτερη παρακολούθηση, υποπτία και πολλά άλλα. Τις προτάσεις σας, τις ε, συστάσεις στο κείμενό σας. Όλα αυτά ήταν πολύ χρήσιμα και εγώ θέλω να υπάρχει ασφαλή δικαίου έτσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότεροι. Α, η κυρία Σαρχεντίνη το είπε. Μας είπε για την αιρεσιμότητα. Τι είπατε. Α, την αιρεσιμότητα σε σχέση με το δημοσιονομικό πλαίσιο, το MFF. Όταν αναφέρθηκε το σχετικό, πανικοβλήθηκαν πολλά κράτη-μέλη. Γιατί θεωρήσανε ότι αυτό θα τις στρίμωχνε, Ιδίω στις χώρες συνοχής. Εμείς θέλουμε αυτό να το συνδέσουμε με οριζόντια χρηματοδότηση, όλου του πόρου πόρους που μοιράζονται στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πώς νοούμε το κράτος δικαίου. Υπό ποιες προϋποθέσεις θέλουμε να ισχύει και άρα να το συνδυάσουμε. Να έχουμε έναν ορισμό περιγραφικό για τη δικαιοσύνη, για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ε, τους εποπτικούς, τους ελεγκτικούς, λοιπόν, και όλα αυτά σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μια περιγραφή, έναν ορισμό πιο αναλυτικό για το πώς βλέπουμε ότι θα πρέπει να ισχύει το δικαίωμα στα κράτη μελή μας, τόσο γίνεται πιο συγκεκριμένο να διασκεδάσουμε τις αμφιβολίες και ε, αυτό να διέπει τους μηχανισμούς λήψη αποφάσεων και έτσι να μοιράζονται οι πόροι κανείς δεν θέλει να πάνε τα πράγματα ανάποδα Γι' αυτό είναι άρα. Τέτοιες αιρεσιμότητες θέλουμε. Και μην ξεχνούμε το όσα ήδη ισχύουν σε την κατανομή των ε, πόρων. Απλούστευση των κανόνων και γι' αυτό και θα πατήσουμε το πόδι στα σπουδαία. Αυτά που μετράνε. Κράτος δικαίου. Για να δούμε τότε τις άλλες ερωτήσεις σας για τη Σλοβακία. Για τη Σλοβακία. Θα δούμε κατά πόσον η υπεξαίρεση των κοινωτικών πόρων ε, βρίσκεται πίσω από αυτή την τραγωδία, από αυτή την αποτρόπια υπόθεση. Όλα αυτά θα τα ελέγξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 2020. Ανεξάρτητη υπηρεσία για τα οικονομικά κακουργήματα στην Ένωση. Είμαι πεπισμένη ότι κάνουμε το σωστό. Και θα ήθελα να καλέσω και άλλα κρατημέλια. Να προσχωρήσει και η Σουηδία, να προσχωρήσει και η Μάλτα, η Πολωνία και η Ουγγαρία σε αυτή την υπόθεση. Καλά. Βέβαια, ελπίζουμε ότι και οι κάτω χώρε θα μπουν στο σύστημα της εισαγγελία. Οπότε προσδοκώνται πάρα πολύ σημαντικοί πόροι, ούτως ώστε να κατανεμηθούν στα σχετικά έργα και για Πολωνία και Ουγγαρία, κατά τη γνώμη μου, ε, θα πρέπει αυτές οι χώρες να το ξανασκεφτούν και το κατά πόσο θα μπουν στην υπόθεση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για την καταπολέμηση της απάτη και της ε, διαφθοράς και είναι κοινή υπόθεση γιατί δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα του αν μας εμπιστεύονται οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Α, τα είδατε. Τι, γίνεται, τι έγινε στη Σλοβακία. Άρα θα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο προς αυτό το μέτωπο και αυτό και εύχομαι και ελπίζω και θέλω ότι αυτοί που διέπραξαν αυτό το αποτρόπιο έγκλημα θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν. Ότι θα μάθουμε το μάθημά μας. Και συγκροτώντας το γραφείο την υπηρεσία των σβάντων της Ευρωπαϊκής Αγγελίας θα παγιώσουμε και αυτές τις αρχές για την αιρεσιμότητα, για τους κοινοτικούς ε, πόρους. Και μπορώ να σας ενημερώσω ότι σήμερα ολοκληρώνουμε τη σχετική πρόταση για την προστασία των καταγγελόντων. Θα είναι οριζοντίου χαρακτήρα αυτή η ρύθμιση και έτσι οι έντιμοι θα έχουν περισσότερες ε, δυνατότητες αν δουν κάτι στραβό ούτω ώστε να το καταγγείλουν και να έχουν την ε, αναγκαία προστασία. Πολύ σημαντικό. Και είχαμε επίσης μια σειρά από ερωτήσεων που όμω δεν ήταν ειδικέ για τον, για τον εισαγγελέα, δεν είχαμε ειδικό θέμα. Για τον γενικό κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα, ναι, υπάρχει προόδος. Ε, σε τρεις κλάδους δουλεύουμε ιδιαίτερως. Προσπαθούμε καταρχάς να συντονίσουμε το έργο για το συντονισμό της νομοθεσίας βεβαίως υπάρχει νομοθεσία αλλά υπάρχει και άλλη συναφής νομοθεσία των κρατών μελών η οποία χρειάζεται επικαιροποίηση. Ως γνωστόν ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Το όνειρό μα για ενοποιημένους κανόνες κινδυνεύει ακριβώς από αυτό, γιατί εκεί υπάρχει το περιθώριο των αποκλήσεων και γι' αυτό επαγρυπνεί ιδιαίτερω η Επιτροπή σε σχέση με ορισμένα κράτη-μέλη μάλιστα ε, και προσπαθούμε σε συνεργασία μαζί τους να τα πείσουμε να μην αποκλίνουν από το πνεύμα και το γράμμα του κανονισμού. Δύο κράτη έχουν προχωρήσει σε υιοθέτηση του κανονισμού, Γερμανία και Αυστρία. κάποια άλλα ολοκληρώνουν τη σχετική δουλειά, ενώ άλλα κράτη-μέλη ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ενσωματώσουν εγκαίρως τη σχετική νομοθεσία. Άρα θα αρχίσει η υλοποίηση του κανονισμού με την απευθείας εφαρμογή, με την άμεση εφαρμογή, χωρίς η εθνική νομοθεσία. που στόχο έχει να αντιμετωπίσει το τα διάφορα κενά στην νομοθεσία, δηλαδή το δημόσιο δίκαιο των κρατών μελών που ενδεχομένως να παρουσιάζουν αποκλείστηση κενά. Αυτά. Ε, Επίση, σε σχέση με ορισμένες επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες ανησυχούν τα μάλα για τους νέους κανόνες. Ε, πολλές από αυτές βέβαια περιτά ανησυχούν γιατί ε, γίνεται η αξιολόγηση κινδύνου για τον ε, τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί ο νέος κανονισμός στις, μικρομεσαίες, στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ε, θα χρειαστούν βέβαια καλύτερες πληροφορίες, συμβουλές. Και αυτό βεβαίως νομίζω ότι είναι δουλειά και των υπηρεσιών προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ε, δεκάδες είναι τα ε, ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνω καθημερινά ερωτήματα των επιχειρήσεων που με ρωτάνε πώς θα εφαρμόσω εγώ την νομοθεσία στην επιχείρησή μου. Απαντώ σε όλα, αν και δεν είναι δουλειά μου. Αλλά πάλι είναι πολύ σοβαρό το θέμα γιατί θα πρέπει αυτός ο κανονισμός ε, στα κράτη-μέλη να ε, διαβάζεται σε συνδυασμό με την εθνική νομοθεσία. Εν πάση περιπτώσει προσφέρουμε την καθοδήγηση, θα συνεχίσουμε και θα επενδύσουμε και άλλα χρήματα στην ευαισθητοποίηση. των επιχειρήσεων και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε ένα ολοκληρωμένο ε, σύστημα και πιστεύω ότι μπορούμε έτσι και να προσφέρουμε τη βοήθειά μας όπως έλεγα για να προετοιμαστούν καλύτερα οι επιχειρήσεις. Ο τρίτος κλάδος δράσης μας έναντι του πολίτη πλέον, γιατί ο γενικός κανονισμός είναι ένα νομοθέτημα βαρύ, με σοβαρές ε, επιπτώσεις αντίκτυπο στην ε, ζωή του πολίτη αλλά και στον ε, δημόσιο τομέα. Αν λοιπόν ο πολίτης δεν ασκήσει, δεν διεκδικήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από το Γενικό Κανονισμό, θα είναι περιττός αυτός θα ματαιωθεί ο λόγος ύπαρξής του και γι' αυτό και θέλουμε να ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση και σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, της ε, τους φορείς προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι αρχές και με τις επιχειρήσεις βεβαίως, γιατί και αυτές θα πρέπει να ενημερώνουν τους ε, πελάτες τους ότι εφαρμόζουν τους νέους κανόνες, γιατί αυτό που ακούω ε, γενικά από τις ε, υπηρεσίες είναι ότι πιστεύουν πως ε, προστασία του προσωπικού βίου των πελατών τους ισοδυναμεί με ενίσχυση της εμπιστοσύνης που τρέφει ο πελάτης αυτούς, σε αυτές. Και πιστεύω ότι έτσι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, όντως θλιβερή ιστορία. Ένα νομοθέτημα πολύ ε, λειτουργικό και χρήσιμο που αποσκοπεί στην ε, καταπολέμηση όλων αυτών των φρικτών περιπτώσεων βίας εις βάρος γυναικών και παιδιών και θα το πω έτσι, με συγχωρείτε πέραν των ε, παραδοσιακών μορφών βίας, λυπάμαι, ελπίζω να μην συνεχιστούν αυτές οι παραδόσεις στην ε, Ευρώπη, αλλά και άλλες μορφές όπως είναι ο ακροτηριασμός των γενετικών οργάνων, η καταναγκαστική γάμη, οι απαγωγές εις βάρος γυναικών και κοριτσιών, δηλαδή πράγματα τα οποία στην Ευρώπη του 21ου αιώνα δεν έπρεπε να έχουν καμία θέση. Και γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια ε, συμμετέσχε ως συμβαλόμενο μέρος στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και ευχαριστώ ιδιαίτερα σε εσά τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μας στηρίξατε σε αυτήν την προσπάθεια. Ιδιαίτερα δεν θέλω να αναφέρω και με συγχωρείτε για την προφορά. Να ευχαριστώ την κυρία Μπονφουά, και την κυρία Κοράτσα Μπίλτ για όλες τις προσπάθειες. Τώρα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή έχουμε επικύρωση από 17 κράτη-μέλη. Κάποια άλλα περιμένουμε ακόμα να προχωρήσουν στην κύρωση, σε κάποια άλλα είναι ε, έχουν ανάψει τα πνεύματα στη συζήτηση. Η Βουλγαρία, παραδείγματι, χωρί να θέλω να καταγγείλω κανέναν, μια και όμω η Βουλγαρία έχει την Προεδρία, είναι καλό να δώσουμε το δικό τους, τη δική του περίπτωση. Παρακολουθώ λοιπόν την, το δημόσιο διάλογο στη Βουλγαρία και διαπιστώνω ότι και ο τίτλο ο ίδιο, Σύμβαση τη Ισταμπούλ, γεννά αρνητικά συναισθήματα. Έχθρα. Δυσκολίες επίσης έχουμε και σε σχέση με τη γλώσσα, τη μετάφραση. Υπάρχει ερμηνεία που λέει ότι με τη σύμβαση αυτή προσπαθούν κάποιοι να φέρουν το τρίτο φύλλο, εκτός του ότι φύλλο και γενετήσια προτίμηση είναι μια αμφιβολή ε, κατάσταση, όχι μόνο στη βουλγαρική αλλά και σε πολλές άλλες γλώσσες. Είναι γλωσσικό το ζήτημα σε μεγάλο βαθμό, σεξ και gender δηλαδή. Άρα λοιπόν ε, έχουμε διάφορα απρόβλεπτα προβλήματα, ομολογώ ότι δεν τα είχα προβλέψει. Επίσης έχουμε έντονες αντιδράσεις από κάποιους κύκλους σημαντικούς και ε, εμπλεκόμενους φορείς που υπενήσονται ότι θα μπορούσε να καταστρέψει την παραδοσιακή οικογένεια η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Εδώ λοιπόν προσπαθώ να εξηγήσω ότι αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε χάρη στη σύμβαση Κωνσταντινούπολης και αυτό το κάνουμε και παντού, δηλαδή προσπαθούμε να απαλείψουμε τη βία εις βάρος των γυναικών, των παιδιών, την ενδοοικογενειακή βία που είναι ένα φαινόμενο εκτεταμένο σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε την κύρωση της συνθήκης. Υπάρχουν κράτη-μέλη της σύμβασης, υπάρχουν λοιπόν κράτη-μέλη, Σλοβακία, επί παραδείγματι, που φαίνεται πως ε, δεν σκοπεύουν να κυρώσουν, αλλά κάποια στοιχεία της σύμβασης ε, μπορούν να τα ενσωματώσουν, από ό,τι φαίνεται, στο ποινικό τους δίκαιο. Προσπαθώ να τους πείσω να κυρώσουν. Ε αλλά αν όχι, αυτή η ε, εναλλακτική δεύτερη λύση που δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά σας το λέω γιατί διαπιστώνω ότι κάποια κράτη-μέλη προσπαθούν έστω κάποια λύση να βρουν. Αλλά τι να κάνω, ε, όσο και αν δεν μου αρέσει, τα κράτη-μέλη αποφασίζουν. Η Ρωμά. Άλλη πονεμένη ιστορία πρέπει να πω. Υπάρχει στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα κράτη-μέλη, εκατομμύρια λέξεις, εκατομμύρια σελίδες, αποτελέσματα μηδέν και γι' αυτό θέλουμε να προχωρήσουμε σε μια πραγματική αξιολόγηση της στρατηγικής για τους Ρωμά σε ευρωπαϊκό επίπεδο Έχω συναντηθεί με τους αρμόδιους για την αξιολόγηση και τους ε, κάλεσα να μας παρουσιάσουν την αληθινή εικόνα και να ε, ε, αξιολογήσουν τι φέρνει αποτελέσματα και τι δεν φέρνει. Ένα παράδειγμα. των περιπτώσεων όπου έχουμε παραβιάσεις λόγω προβλημάτων στην ε, προσφερόμενη ε, στα παιδιά των Ρωμά εκπαίδευση και βεβαίως θα σας πω ότι θα συνεχίσουμε αυτές τις διαδικασίες σε παραβάση αλλά θα προτιμούσα να δω πραγματικά αποτελέσματα και αποτέλεσμα για μένα είναι η ουσιαστική αλλαγή όχι μόνο η εισαγωγή της νομοθεσίας. Άρα λοιπόν σε ανάλυση της κατάστασης με ορισμένα κράτη-μέλη και σε επικοινωνία και συνομιλίες με δασκάλους, σε σχολεία, συνομιλίες με γονείς, ε, με ε, ακτιβιστές, πολιτικούς, διαπιστώνω ότι το πρόβλημα από μόνο του δεν λύνεται. Μπορεί να υπάρχει η νομοθεσία σχετική με την ε, προσφερόμενη ε, δημόσια εκπαίδευση παραδείγματι στα κράτη που αποκλείει, που απαγορεύει τις διακρίσεις αλλά πρέπει και σε συνεργασία με τους γονείς να εργαστούμε και να καταπολεμήσουμε την ανεργία, τη φτώχεια τη διακριτική μεταχείριση και όχι μόνο στην εκπαίδευση. Αυτό είναι μια δουλειά που σημαίνει ότι πρέπει να εμπλακούν όλοι οι φορείς σε όλα τα κράτη-μέλη και μπορεί να είναι κλεισέ και δεν μου αρέσει καθόλου ο όρος ολιστική προσέγγιση, αλλά εν προκειμένου είναι εύστοχη και τι χρειαζόμαστε. Θα επισκέπτομαι λοιπόν πάντα τις χώρες αυτές όπου υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή του στρατηγικής για τους Ρωμά και στη διάρκεια του έτους θα συνεχίσω γιατί προσπαθώ να αντιληφθώ ποια είναι τα προβλήματα που προκύπτουν και ε, θέλω να κοιτάξουμε ε, προβλήματα και λύσεις εκεί όπου αυτές έχουν φέρει αποτελέσματα διότι θα, αρχίσουμε, θα έρθει η ώρα βέβαια να συζητήσουμε συγκεκριμένες προτεραιότητες για ένα πλαίσιο δημοσιονομικό, ε, για την δημοσιονομικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να αποφύγουμε τα προβλήματα του παρελθόντος. Πρέπει λοιπόν να είναι πιο στοχευμένα τα κονδύλια που θα διατίθενται. Για τους Ρωμά λοιπόν αυτό για τις διακρίσεις αλλά και για την ε, ε, αφρικανοφοβία και άλλα θέματα. Η Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί για να καταστήσει απολύτως σαφές ότι είναι αφόρητη και ανυπόφερη η, η αδίποτε διάκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε στρατηγική για την ξενοφοβία που πρέπει να υλοποιείται σε κάθε κράτος μέλος. Έχουμε μια σειρά από ε, νομοθετήματα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και πρέπει να ε, προωθήσουμε στην υιοθέ, την υιοθέτηση της οδηγίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων για την ίση μεταχείριση. Τώρα μας ρωτάτε τι γίνεται εδώ. Ε, λοιπόν, όντως το Συμβούλιο έχει παρεμποδιστεί η ε, εξέλιξη του θέματος. Θέλω να κάνουμε τη συζήτηση με τους υπουργούς εφέτος και ε, περιμένω να ακούσω επιχειρήματα ότι θα κοστίσει ακριβά και όλα αυτά. Και θέλω να επικαιροποιήσω τα οικονομικά στοιχεία που έχουμε, γιατί έχουμε νομοθεσία με στοιχεία του 2008 ε, αντιλαμβάνομαι βεβαίως ότι αν δεν υπάρχουν ενημερωμένα στοιχεία, ανάλυση, αξιολόγηση συνεπειών, δεν είναι δυνατόν να προβάλλουμε και το αντιεπιχείρημα ότι ναι μπορεί να σας κοστίσει, αλλά τα ωφέλη και σε οικονομικούς όρους είναι αυτά και αυτά. Ε, και θα ήθελα βεβαίως να αφιερώσω ε, πολύ ενεργητικότητα σε αυτό το θέμα και φέτος θα σας ενημερώσω για το πώς ε, ε, προχωρεί η συζήτηση στο Συμβούλιο ε, και στο δεύτερο εξάμεινο. Υπάρχει επιλογή της ενισχυμένης συνεργασίας, αλλά για μένα δεν είναι πραγματική επιλογή, γιατί σημαίνει ότι μόνο κάποια μπορούν, μπορεί να δεχθούν να συμμετάσχουν. Για τον κύριο Γιούρεκ δεν έδωσε απάντηση. Άμεση δημοκρατία, ναι. Να σας πω ποια είναι η προσωπική μου γνώμη. Δεν έχω καμιά αντίρρηση για την, προσωπική, για την άμεση δημοκρατία και τα δημοψηφίσματα πάντα όμως πρέπει να κοιτάμε και τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό. Διδάγματα μπορούμε να αντιλούσουμε φερρυπίν από το Brexit. Γιατί είναι εύκολο να γίνει πλησία κεφάλου και να επηρεαστούν ε, οι πολίτες με ψευδείς ειδήσει. Είναι απίστευτο το πόσο εύκολο είναι. Και πιστεύω ότι πρέπει όλες τις ε, συνθήκες αλλά και ε, τις περιστάσεις από τις οποίες διαξαγόνται τα δημοψηφίσματα να τις εξετάσουμε με μεγάλη σοβαρότητα. Βέβαια τα κράτη-μέλη αποφασίζουν, αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν τις υπεύθυνε αποφάσεις και σε εκ τούτου δεν μπορώ να δώσω για θέματα που αφορούν τα κράτη-μέλη δεν μπορώ να εκφράσω επίσημα θέση. Για το θέμα του Γενικού Γραμματέα σας ευχαριστώ για την ερώτηση, με ξαφνιάσατε, δεν την περίμενα, η κυρία Εντφέλτ που πάντα έχει εύστοχες ερωτήσεις. Οφείλω να πω ότι δεν έχω λάβει από τους ε, ε, πολίτες που συχνά μου αποστέλνουν επιστολές για τη φτώχεια, τη διακρίση, ε, την εγκληματικότητα, επιστολές. Από αυτούς λοιπόν τους πολίτες δεν έχω λάβει καμία σχετική ερώτηση. Η Επιτροπή ως λογικό όργανο ε, ενέκρινε την, ε, τον διορισμό και τίποτε περισσότερο δεν έχω να σας πω. Αλλά βλέπετε ότι δεν απέφυγα την ερώτησή σας. Ξέχασα κάτι μήπως. προστασία προσωπικών δεδομένων ε, στα ε, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ως Επιτροπή ε, εντατικά εργαζόμαστε για την ε, απεμπλοκή του θέματος. Θέλουμε μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός, ε, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, να είμαστε απολύτως έτοιμοι. Έχουμε βρει, πιστεύω, πολύ καλές λύσεις και για τις υπηρεσίες ε, επιβολής και παρακολούθησης της ε, ε, εφαρμογής νομοθεσίας, γιατί οπωσδήποτε το χρειαζόμαστε αυτό. Επίσης για την ηλεκτρονική προστασία για την προσωπικά δεδομένα στο, στο ηλεκτρονικό πεδίο, το ίδιο. Και επίσης, τι άλλο θέλατε να ρωτήσετε την κυρία Γιώργο. Equal Treatment Directive. Α, ναι, για την ίση μεταχείριση και την οδηγία. Ε, το είπα ότι για φέτος προβλέπουμε η συζήτηση που θα θίξει την ε, πραγματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί θα μας αποσχολήσει, αλλά δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική αλλαγή μετά την πιο πρόσφατη συζήτηση. Οπότε από την Άνοιξη θέλουμε να δούμε τους ε, αριθμούς και τους μακροοικονομικούς όρους, να εκτιμήσουμε καλύτερα το κόστος και τα ωφέλη και θα επανέλθουμε στο θέμα ξανά το φθινόπωρο. Ελπίζω, ελπίζω ότι η ενισχυμένη συνεργασία δεν θα μας προδώσει. Ε, δεν θα είναι η λύση για το θέμα αυτό. Δεν θα είναι η μόνιμη εναλλακτική. Αλλά από αυτά που άκουσα από την τελευταία φορά από τους υπουργού είναι βασικό θέμα και πρέπει όλοι να συμμετάσχουμε για την οδηγία της ίσης μεταχείρισης δεν ανήκει. Μάλλον υπάγεται σε ένα συγκεκριμένο Υπουργείο στα κατημέλη, αλλά χρειάζεται συνεργασία και άλλων Υπουργείων. Αυτό είναι ένα θέμα οριζόντιο. Οπότε γίνεται ακόμη πιο δύσκολο σε επίπεδο κάποιων κατομελών. Και για την εμπορία των ανθρώπων δεν έχω τέτοιες πληροφορίες. Λυπούμε. Μπορώ αν θέλετε να σας απαντήσω γραπτός. Ευχαριστούμε. Ήταν μαραθώνια η απάντησή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις τόσο διεξοδικές τους ερωτήσεις. Ήταν τόσο διαφερμένος ο διάλογος που πιάσαμε και το κάθε παραμικρό σημείο του χαρτοφυλακίου σας. Σε μερικούς μήνες ελπίζουμε ότι θα έχουμε και τα απαραίτητα στοιχεία. Ναι, ε, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ευχαριστώ πολύ για τι ερωτήσει σα και είμαι στη διάθεσή σα για τη μελλοντική μα συνεργασία. Ε, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που να συζητήσουμε. Σα ευχαριστούμε πολύ, σα ευχαριστούμε και για τη δουλειά σα. Συνάδελφοι, σα ευχαριστώ όλου. Το τελευταίο σημείο να βάλετε. Πάμε απευθείας στη συνεδρία των συντονιστών.